Ψηφίζουμε. Τροπολογία 68. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος κατά. Αποχές απορρίπτεται. 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 69. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πηγαίνουμε λοιπόν τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 79. Υπέρ. Κατά άποχες απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά άποχες απορρίπτεται. Τροπολογία 4. 81, ήτρε 14, τραν 9, είναι παρόμοιες. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Άποχες. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 84. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Χωριστή ψηφοφορία για την Ενοποιημένη τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Θα το κοιτάξουμε ηλεκτρονικά. Κανείς δεν ψήφισε με το χέρι. Άρχεται η ψηφοφορία. Επαναλαμβάνω. Ψηφίζουμε τώρα στην προσθήκη στην ενοποιημένη τροπολογία 3 στη σελίδα 4 στο κειμενό μου. Ψηφίσατε όλοι. Οι πράσινοι έχουν μία ψήφο παραπάνω. Υπάρχουν ασάφειες. Ξανά, ξανά. Ψηφίσαμε μόλις τώρα την ενοποιημένη τροπολογία 3 και πρέπει να κάνουμε μια χωριστή ψηφοφορία για το τραπεζικό σύστημα. Λοιπόν, ξεχωριστή ψηφοφορία. Οι συγητής και οι συγητές συμφώνησαν λοιπόν για αυτό το τραπεζικό σύστημα και αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε ηλεκτρονικά, διότι κανένας από εσά δεν σήκωσε το χέρι του. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λοιπόν, Τρεις συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Αν θέλετε, παρακαλώ, ευπρόσδεκτοι είστε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 39 ψήφους κατά και 20 υπέρ. Πήδαμε λοιπόν σε μια ξεχωριστή λίστα ψηφοφορίας. Για, σε μένα είναι η σελίδα 24, η τελευταία. Τη βρήκατε όλοι? Είστε έτοιμοι? Στο τέλος λοιπόν του δικού μου καταλόγου υπάρχει μια ξεχωριστή ψηφοφορία. Είστε σε θέση όλοι να ψηφίσετε. Πείτε. Ναι. 85. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Όχι, όχι, θα το κοιτάξουμε και αυτό ηλεκτρονικά. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας. ...32 ψήφοι Περεγκρίνεται. Όλα τα υπόλοιπα καταπίπτουν. Επιστρέφουμε τώρα... ...στη σελίδα 7 ψηφίζουμε την Ήτρε 17. Σας περιμένω μέχρι να βρείτε που είμαστε. Ήτρε 17. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 114. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δύο όμοιες τροπολογίες, 117 και τραν, Ποιο είναι υπέρ, τραν 12, ποιος είναι κατά, Αποχές εγκρίνονται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην 118 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές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 αποχές εγκρίνεται. 111. Με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 και ήτρε 20 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήτρα 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 133. Υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 133 ηλεκτρονικά. 133 ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε. Το ΕΛΚ έχει δύο παραπάνω. Δύο ψήφους παραπάνω. Μία ψήφο παραπάνω. Τώρα, μάλιστα, πέρας ψηφοφορίας, 44 υπέρ 21 κατά εγκρίνεται. 134 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 138 και τραν 16 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ας κοιτάξουμε ηλεκτρονικά όμως, τραν 16 και 138. Ψηφίσατε. ΕΛΚ. Πάλι μία ψήφος παραπάνω. Τώρα είμαστε εντάξει. 27 υπέρ, 37 κατά, απορρίπτεται. Ήτρα 24 υπέρ, Κατά. Αποχές. Κοιτάζουμε ηλεκτρονικά. Ήτρα 24. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στη σελίδα 14, τροπολογία 152. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 153. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρα 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρε 27 και τραν 18. Θα ψηφίσουμε και τις δύο μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 157. Καταπίπτει 157. 167. εξήντα επτά στη σελίδα 16. Ποιος είναι υπέρ. Εκατόν 67. Σαμπίνε βίλς στη σελίδα 16. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 166, 168 και 170. Θα τις ψηφίσουμε μαζί. Είναι ομοίες ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 169. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 175 υπέρ, κατά, Εγκρίνεται, αλλά θα κοιτάξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. 175. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τραν 21 καταπίπτει και 22 καταπίπτει. Πάμε λοιπόν στην 176 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 177 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, Τιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 1 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνατε. 28 και 29 είναι παρόμοιες. και είναι υπέρ. Κατά. Θα κοιτάξουμε ηλεκτρονικά 28 και 29. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε. ΕΛΚ. Μία ψήφος παραπάνω. Μάλιστα, ήρθαν τα πράγματα στη θέση τους τώρα. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτονται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρε 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 33 και τραν 2. Μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Η 34 καταπίπτει. Ψηφίζουμε την τροπολογία 1, 35, ποιος είναι υπέρ, ποιος κατά, αποχές, δεν είναι σαφέ. Θα το κοιτάξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 1, 35, 33 και 35. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα, Εγκρίνονται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 49 ήτρε 8 ήτρε 49 και ήτρε 8. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Ήτρε 7 υπέρ κατά, άποχες, εγκρίνεται. 50 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά, Αποχές απορρίπτεται. Μάλιστα, κάνουμε άλλο ένα άλμα στην τροπολογία 3 και στην ήτρε 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 11. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 66. Υπέρ. Κατά αποχές, απορρίπτεται. τράνεπτα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στην πρώτη οριστική ψηφοφορία για την πρόταση ή ηλεκτρονικά όπως πάντα. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται 45 ναι, 15 όχι, 3 αποχές. Πάμε τώρα στην οριστική ψηφοφορία για το σχέδιο θετικού ψηφίσματος ως σύνολο. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ζητώ λοιπόν από τον εισηγητή εάν... Ναι, θέλει, θέλει, μου λέει. Κρίς. Να μας πείτε, λίγο τις ψήφους για αυτή την ψηφοφορία. Τελευταία. 47 υπέρ. 17 κατά. Μία εποχή. Στη δεύτερη. Και τώρα. Για την εντολή και ξέρω ακριβώς το νούμερο, 35 χρειαζόμαστε. 35 ψήφους και γι' αυτό χρειάζεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για την χορηγήση της εντολής. Ψήφισαν οι πάντες. Πέρασε η Κύριε Ρέμερ, έχετε λάβει εντολή και σας ζηλεύω, σας φωνώ.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 και προχωράμε σιγά σιγά από τα πιο απλά στα πιο δύσκολα. Μπορούμε να έχουμε λίγη ησυχία παρακαλώ. Όσοι συνάδελφοι δεν θέλουν να παραμείνουν για την ψηφοφορία, παρακαλώ ησύχως να αποχωρήσουν. και οι σκιώδεις ηγητές για τα οχήματα παρακαλούνται έξω από την πόρτα να κάνουν τι πραγματεύσεις τους. Και έτσι μπορώ να ξεκινήσω με την έκθεση του συναδέλφου Φράνκο, 7ο πρόγραμμα πλάσ, δράσεως. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, απορρίπτεται. 107. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 108 υπέρ κατά άποχες απερίφθη 110 υπέρ κατά απορρίπτεται 109 υπέρ κατά άποχες απερίπτεται 111 όχι θα επαληθεύσουμε την 111. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Ψήφισαν όλοι. Όχι, με συγχωρείτε. Ε, παραλαμβάνω, 109 λέει ο πρόεδρος τώρα. 109, την 109 παραληθεύουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 111 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 7. Υπέρ. Θέλετε να επαληθεύσουμε. 119 λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 7 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 120 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 100. Ε, άγκρη πρώτη της ε, Γεωργικής υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 124 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 123 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 125 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δύο της Γεωργίας υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 127 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη 128 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 129 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Την 130, αυτή θέλετε να απολυτεύσουμε. Ευχαριστώ. 130. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά την 130. Πέρας στις ψηφοφορίες. Ναι, τι να σας πω. 131 τώρα λοιπόν. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 132 υπέρ. Κατά σε απορρίπτεται. 133 υπέρ. Να επαληθεύσουμε. 132. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. <laughs> Να έχετε εμπιστοσύνη στον πρόεδρο, απορρίφη. 133. Υπέρ. Κατά. Αποχέσα, 8 σε δύο τμήματα. Πρώτο παρακαλώ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 134 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Γεωργική 3 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Το δεύτερο τμήμα, όχι, δεν έχει λόγο να ψηφιστεί και έτσι πάμε στην 135 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται, 136 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, 137 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθεται, 138 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, 139 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Την 9 πάλι λοιπόν. Υπέρ. Ξαναψηφίζουμε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της ε, τροπολογίας 4 της Γιώργης Κατά. Αποχές απερίφθη. Στην 140 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 142 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές περιφθεί. Επαληθεύουμε. 146 ε, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τις ψηφοφορίες. Για μια ψήφο εκκρίνεται. Καλά κάναμε και το επαληθεύσαμε λοιπόν. 147 υπέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 148 ψηφίζεται υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη, 149 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη, 152 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη, 153 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη, 154 υπέρ, Α, ναι, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Βιάστηκα, έχει γίνει δεκτό. 154 τώρα, υπέρ. Κατά. Άποχες. Απερίφθη. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 156 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη ενοποιημένη παριθμόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ενοποιημένη 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 15 τώρα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 166 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 165 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 167 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται 168 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 169 δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ. Κατά. εποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. εποχές Απερίφθη. Επαλήθευση. Ευχαριστώ. Εψήφισαν όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Ω, σας ευχαριστώ. Μερσή. Από εδώ φαινόταν διαφορετική η ισορροπία. 170 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα της 170 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 171 δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 173 και 9 της ε, γεωργικής μαζί υπέρ. Κατά. Απερίφθη λέει ο πρόεδρος να επαληθεύσουμε. Ευχαριστώ σαν και φιλελεύθεροι. Μαζί ψήφισαν. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Ε, πρέπει να... Πρέπει να διορθωθώ. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Η 16 τώρα. Τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Το τρίτο τμήμα Πρέπει και αυτό να το ψηφίσουμε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα, η 175 ψηφίστε μαζί με την 11 της γεωργικής υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, επαληθεύουμε τις δύο τροπολογίες, επαληθεύουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίες. Απερίφθη. Απερίφθησαν. 176 πρώτο τμήμα και προφορική τροπολογία στο δεύτερο τμήμα της. Πρώτο τμήμα λοιπόν υπέρ. Κατά. Άποχες. Απερίφθη και άρα καταπίπτει το δεύτερο τμήμα και πάμε στην 178 υπέρ. Κατά. Εποχές απερίφθη. 181 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απερίφθη. Ελέγχουμε την 181 επαλήθευση ηλεκτρονική. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Πότε πότε έχουν και δίκαιο οι φιλελεύθεροι. Απερίφθη. Καταπίπτει 177, 179 τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 180 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά την 180. Ψήφισαν όλοι. Έγκρινεται. 182. Όχι, με συγχωρείτε λέει ο πρόεδρος, στη 12 της Γεωργίας, σε τρία τμήματα. Πρώτο παρακαλώ. Κατά αποχές απερίφθη. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Πρώτο. Θα επαληθεύσουμε το πρώτο, μάλιστα. Η ηλεκτρονική επαληθεύση. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Δεύτερο τμήμα. Πάλι ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 183 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 184 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 185 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 188 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 187 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 189 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 190 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 191 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 192 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα 192 ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν οι πάντες πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 193 υπέρ Κατά. Αποχές απερίφθη 194 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 197 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Αλλά σκάνουμε για μια φορά την ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψήφισαν οι πάντες. Πέρα τις ψηφοφορίες. Απερίφθηκε λίγο. 195 μαζί με την 13 της Άγκρη υπέρ, κατά αποχές. Απερίφθη 196 υπέρ, κατά αποχές. Απερίφθη 199 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. 198 μαζί με την 14η της για γιατί να ταυτόσουμε, υπέρ, κατά. Αποχές. Απερίφθη. Σαν. 19 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 19 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 15 της Γεωργίας υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 20 υπέρ. Α, 200 λέει ο πρόεδρος, με συγχωρείτε. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 201 καταπίπτει. 16 της Γεωργίας υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 202 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 204 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 205 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 207 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 206 πίπτη. 208 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 17 της Γεωργικής, δύο τμήματα. Πρώτο παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Όχι το δεύτερο τμήμα γιατί έχει καταπέσει. Πάμε στην 109 λέει ο πρόεδρος. 209 πρώτο τμήμα σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. Και επαληθεύουμε τη 209 πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα στην κατατμήματη ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά ψήφισαν όλοι. Δεύτερο τμήμα της 209. Στη 209, πρώτο τμήμα, δεύτερο τμήμα στα κατατμήματα. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απερίφθη. 209, δεύτερο τμήμα, σε δύο τμήματα, σε δύο κομμάτια και ψηφίζουμε το πρώτο υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 210 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 211 και 12 μαζί υπέρ κατά άποχες απερίφθη 213 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 214 υπέρ κατά άποχες απερίφθη 215 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη 216 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 217 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 16 της 18 της Γεωργίας υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκριν. Απερίφθη 22 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 218 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 219 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 24 πρώτο τμήμα Πρώτο τμήμα, μία ψηφοφορία ενιαία. Υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 24 δεύτερο τμήμα. Σε τέσσερα κομμάτια, τέσσερα τμήματα. Είναι μια ψηφοφορια ενιαια υπερ κατα 24 όλο αυτό. Ε, ας ψηφίσουμε λοιπόν υπέρ. Να το επαναλάβω. Ωραία, λοιπόν. Τροπολογία 24. Δεύτερο τμήμα. Second part. Και από εκεί το δεύτερο τμήμα, το second part πάλι. Του δεύτερου τμήματος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το υπόλοιπο. Καταπίπτει. Και πάμε στην 25. Υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Κάποιος μου δώσε ένα χαρτάκι ότι θα μας φέρουν καφέ σε λίγο ή και τσαγάκι αν θέλετε. Για το ημίχρονο ξέρετε. 220 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 221 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 222 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 223. επαληθεύουμε τη 222. Ψήφισαν όλοι. Το ΕΛΚ έχει έναν περισσευόμενο. Εγκρίνεται. 223 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ε, παληθεύουμε καλύτερα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. 224 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν απορρίπτεται, δεν είμαι σίγουρος. Ας την ξαναψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 225 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 226 πρώτο τμήμα. Πάλι έχουμε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα λοιπόν της 226 πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα του πρώτου τμήματος υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 226 δεύτερο τμήμα και πάλι σε τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σε φες ηλεκτρονικά παρακαλώ το δεύτερο τμήμα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Διακόσια υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 228 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 27. 27. Με μια προφορική τροπολογία παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 229. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά αποχές απεριφθεί. Ενοποιημένη 4 υπέρ. Κατά αποχές συγκρίνεται 236 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. «241 παρακαλώ υπέρ, κατά αποχές απερίφθη, 21 της υπέρ, κατά αποχές απερίφθη, ενοποιημένη 5 υπέρ, κατά Αποχές. Εγκρίνεται. 245 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 247 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 248 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 251 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 249 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 33 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ Κατά. Αποχές δεν ναι, είναι σαφές. Το δεύτερο τμήμα του 33 παρακαλώ, ηλεκτρονικά, ψηφίσατε όλοι, πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 250 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 22 της Αγιοργικής υπέρ, κατά αποχές απερίφθη 252 υπέρ κατά αποχές δεν είναι το αποτέλεσμα Επαληθεύουμε τη 252 ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Μου λένε ότι οι φιλελεύθεροι ψήφισαν λάθος. Ε, ήταν σαφές. 250, 252, αυτήν ψηφίζουμε. Ξανά. Ψηφίζουμε τη 252 ηλεκτρονικά. Ναι, άμα δεν θέλετε, και είναι πρόβλημα των φιλελεύθερων, θα στο πούμε ότι είναι πρόβλημα των φιλελεύθερων και ας προχωρήσουμε. 253, δεν έχω καμία όρεξη. 253, ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 255, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 256 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 257 υπέρ. Κατά. Αποφε... Αποχές. Απορρίπτεται. 258 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 259 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 260 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται 261 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μάλιστα, προχωράμε. Κάνουμε ένα άλμα στη σελίδα 28. 276 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται ή όχι. 2, 2,76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2,73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 274 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 275 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αγαπητέ συνάδελφε, αν σας ενοχλούμε την ώρα που μιλάτε στο τηλέφωνο, πείτε μας, εντάξει, μην σας διακόπτουμε. Άγκρι 23, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 2,78 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 277 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 279 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 280 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Ενοποιημένη τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 284 σε δύο μέρη, πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές και αυτή εγκρίνεται. 286 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 287 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 288 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 14 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2,98 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2,99 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 300 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άγκρι 24 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 301 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 402 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 303 καταπίπτει, ενωπημένη 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 308 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ενοποιημένη 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 318 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται ενοποιημένη 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 39 χωριστή ψηφοφορία πρώτο μέρος υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές δεν είναι σαφές επαληθεύουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο μέρος της 39. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. εγκρίνατε. 325 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 326 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 327 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 332 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 328 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 329 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 330 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 3.31 υπέρ. Συγγνώμη, σε δύο μέρη, 3.31 το πρώτο μέρος υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 333 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται 335 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 334 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 336 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 3.37 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 3.38 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 339 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 340 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Άγκρι 25 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 341 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 342 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 363 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 364 κατά πάμε στην 343 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 344. Όχι. 343 απαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 3.44 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 3.45 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Μάλιστα, ημίχρονο. 3.46 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3.47 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3.49 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 3.48 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.50 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 351 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 352 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 353 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 355 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 354 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 356 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Άποχες. Να δούμε ηλεκτρονικά. 42. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται. Ενοποιημένη 11. Υπέρ. Κατά. Αποχής εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 361 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 362 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 365 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 366 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 367 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 368. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 369. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 370. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 371 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 372 υπέρ, κατά, Δεν είναι σαφές, θα επαληθεύσουμε. 372. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Φιλελεύθερη. Ένας περισσεύει. Μία ψυχός περισσεύει. Μάλιστα. 60 υπέρ. Είτε ήμουν πολύ γρήγορος είτε ήμουν πολύ αργός. Είναι σαφέστατο όμως εγκρίνεται. 473 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 26 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 374 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 375 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε. 375 ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 376 πίπτη, 377 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 378 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 379 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε. Ηλεκτρονικά. Μόνο 10% από σας ψηφίσατε. ηλεκτρονική επαλήθευση, τροπολογία 50. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. 380 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 381 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 51. Χωριστή ψηφοφορία σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 384. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 385. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 386. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άγκρι 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άγκρι 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 388 έχει αποσυρθεί. 387 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 389 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 391 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 393 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 394 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 395 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 396 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μάλιστα 397 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ενοποιημένη 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 402 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 403 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 404 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 405 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 406 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 407 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 408 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 412 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 409 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 410 και 11 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ναι εγκρίνεται 413 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 414 415 καταπίπτουν αυτές οι δύο 416-418 ταυτόσημες υπέρ Συγγνώμη, 417 ψηφίζουμε. Παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 416 και 18 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Θα ε, πας επαληθεύσουμε όμως. 4-16-4-18. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 4-19. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άγκρη 29. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 420 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 421 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 422 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 423 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4-24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 426 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 428 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 429 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 430 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 431 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 4.32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 433. Χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Θέλουμε να επαληθεύσουμε τώρα την 433 πρώτο μέρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απίστευτο. Οι σοσιαλιστές έχουν μια ψήφο παραπάνω. Αλλά ποτέ δεν είναι αρκετή. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. Δεύτερο μέρος της 433. Ποιος υπέρ, κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές, επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε. Πέρασε. Απορρίφθηκε. 54, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4.34. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 53. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 4.35. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 4.36. Υπέρ. Είμαι αλλεργικό σε λίστε ψηφοφορία πάνω από 50 σελίδε, λέει ο συνάδελφο. Ποιο είναι υπέρ, λοιπόν. Κατά. Απορρίπτεται. 4.37. Υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. 4.38. Υπέρ. Κατά. αποχέ, απορρίπτεται. 4.39. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4.40. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 31 υπέρ κατά όχι κατά Κατά πίπτη και αυτή και αυτή. 4.42 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 443 καταπίπτει. 444. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 445. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Άγκρι 33 υπέρ. Κατά Αποχέ. απορρίπτεται. Άγκρι 34 υπέρ. Κατά Αποχέ. απορρίπτεται. 446 υπέρ. Κατά απόχέ, απορρίπτεται. Άγκρι 35 υπέρ. Κατά αποχέ, απορρίπτεται. 447 υπέρ. Κατά Αποχέ. εγκρίνεται. 448 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Άγκρι 36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Α, συγγνώμη, είναι ταυτόσιμε. Λέει να τις ψηφίσουμε μαζί 448 και άγκρι 36. Απορρίφθηκαν και οι δύο. 449. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 450 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 453 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρις 37 υπέρ. Επαλήθευση της 453. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Άγκρι 37. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 451. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 454 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 455 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 456 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 457 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 458 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4,59 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ. 62 εγκρίνεται. Ναι, 62 εγκρίνεται. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Τα είπα λάθος. 64 υπέρ. Κατά. Α, εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 460 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 461 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 63 πίπτη. Πάμε στην 4... 62 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 464 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 465 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 467 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 468 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 67 σε δύο μέρη. Το πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές να το απαληθεύσουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. 469 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 470 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 471 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4,72 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4,73 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται.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 Εγκρίνεται 4,85 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 4,86 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4,87 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 4,88 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 4,89 υπέρ. Κατά. Υπέρ. Εγκρίνεται εποχή εγκρίνεται. Το 70 καταπίπτει, 490 καταπίπτει, 491 υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. 492 υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 493 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 494 υπέρ. Κατά. απόχέ. εγκρίνεται. Απορρίπτεται. 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4,95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4,96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4,97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4,98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4,99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 500 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 501 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 502 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 503 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πάμε στα εξατηλογικές σκέψει. 76. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 77. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συγγνώμη, εγκρίνεται. 2. Τοπολογία υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 78. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίθηκε ομόφωνα λοιπόν και αυτό. Καμία, κανένα συμβιβασμός. 79 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 82 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 83 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται 94 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 95 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 96 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται 97 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 97. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Να περιμένουμε λοιπόν. Τώρα ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 80. 98. Τροπολογία 98. Ναι. Περδέψαμε τις σελίδες. Τροπολογία 98. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 100 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση στην 101, έρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται. 102. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 104. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Το πρώτο μέρος ήταν αυτό. Οριστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πρώτη ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται 46 ψήφους υπέρ. Τώρα ψηφίζουμε το ψήφισμα στο συνολό του. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται μεγάλη ψηφοφορία. Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω τον εισηγητή, κύριε Φράγκο. Θα ήθελα να σας πω συγχαρητήρια. Μεγάλη στήριξη προς το πρόσωπό σας. Να σας ρωτήσω εάν θέλετε να λάβετε διαπραγματευτική εντολή από αυτήν την Επιτροπή. Ναι, βλέπω πως θέλετε, ουί μου λέτε. Μάλιστα, οπότε ψηφίζουμε για τον κανόνα 70 για την ε, ανάθεση διαπραγματευτικής εντολής. Χρειαζόμαστε 35 ψήφους για να πραγματοποιηθεί. Ψηφίσατε. Πέρας. 48 ψήφοι υπέρ, 7 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια. Η εντολή είναι ολοδική σας, αγαπητέ συναδέλφοι Φράγκο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να ευχαριστώ θερμά και ειλικρινά όλους τους συναδέλφους οι οποίοι μου έδωσαν αυτή τη διαπραγματευτική εντολή. Σκοπεύω να συνεργαστώ όσο πιο στενά μπορώ με την Ιρλανδική Προεδρία για ένα φιλόδοξο, αποτελεσματικό και ρεαλιστικό έργο. Ευχαριστώ τις πολιτικές ομάδες, τους συναδέλφους, το προσωπικό τους για όλη τη συνεργασία και την υποστήριξη, όλο το προσωπικό που στήριξε εμένα, τη δική μου ομάδα που με τόση εφοσίωση όλους αυτούς τους μήνες μου συμπαραστάθηκε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Φράγκο. Α, θέλει και ο κύριος Γιολάινεν το λόγο. Ένα μόνο πράγμα συγχαρητήρια στον εισηγητή και συγχαρητήρια ε, και ευχαριστίες μάλλον για την πολύ συνεργατική του στάση αυτή την έκθεση για το 7ο πρόγραμμα δράσεως. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι νομίζω μπορούν να συμφωνήσουν σε αυτό. So, ich bitte doch diejenigen, die jetzt. Θέλω να ζητήσω λοιπόν τώρα από εκείνους οι οποίοι δεν θέλουν να συμμετέχουν στις συζητήσεις για τον καπνό να κάνουν ησυχία. Ο κύριος Σούλμερ. Θα ήθελα να ρωτήσω πρόεδρο. Είναι ρεαλιστικό έχουμε καμία πιθανότητα το τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης να το συζητήσουμε ή θα αναβληθεί για την προσεχή φορά. Η ψηφοφορία έχει αναβληθεί. Άρα δεν μας πιέζει τίποτα. Ο πρόεδρος. Ναι. Θα, θα αξιοποιήσουμε το χρόνο που χρειάζεται για το καπνό. Γιατί είναι από τα σημαντικά νομοθετήματα της τρέχουσας Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι μας επιτρέπει ο χρόνος. Προτιμώ να το αφήσουμε πρόεδρο τότε. Ε, θεωρητικά ναι, μπορούμε να το αναβάλουμε. Κύριε Ούλμερ, θέλετε να το αφήσουμε. Καλώς. Ο κύριος Φιέλνερ. No, no, just eager to get started. να ξεκινήσουμε. Καλώς. Έχουμε και την εισηγήτρια, λοιπόν. Να ακούσουμε τις ε, παρεμβάσεις με την κυρία Μακάβων πρώτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ που μου το λόγο. Κατά τη συζήτηση που κάναμε πριν να σας παρουσιάσω το σχέδιο έκθεση, είχα πει ότι σε γενικές γραμμές υποστηρίζω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσέγγιση που ακολουθεί για την επανεξέταση νομοθεσίας για τα προϊόντα καπνού. Έχουμε κάνει πολλά στην Ευρώπη, αλλά όχι αρκετά ακόμη. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν νέε τακτικέ ε, που έχουν σκοπό ουσιαστικά να αγκαλιάσουν, να στρατολογήσουν νέου καπνιστέ, νέε γενιέ καπνιστών. Αυτό προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτή την οδηγία. Και θέλω να σα υπενθυμίσω, συναδελφοί, όσοι ήταν παρόντε την προηγούμενη φορά, μετά την αναθεώρηση του 2001, από τότε και μετά, όλε οι χώρε τη Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσυπέγραψαν την περίφημη σύμβαση πλαίσιο κατά τον του καπνού, την FCTC, με στόχο την αντιμετώπιση της χρήσης ε, του καπνού και την αντιμετώπιση του φαινομένου της δημιουργίας των καπνιστών. Το είπα και τελευταία φορά και το ξαναπώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ηγείται παγκοσμίω στον έλεγχο ε, του καπνού. Έχουμε πολλούς καπνιστές, περισσότερους από πολλά, αλλά μέρη του κόσμου στις έχουν 18,1%, ο Καναδάς 17%, η Βραζιλία 15%, εμείς κατά μέσο όρο 28 με 29% των νέων μας συνεχίζουν να είναι καπνιστές και από ό,τι ακούμε η πλειοψηφία των νέων ξεκινούν από παιδιά ε, να καπνίζουν. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να αναλάβουμε δράση για να σταματήσουμε αυτό το φαινόμενο όσο μπορούμε. Λοιπόν, οι βασικές προτάσεις που κάνει η Επιτροπή στην πρώτη οδηγία είναι καλές προτάσεις, απλά θέλω να διατρέξω ε, τα σημεία που εγώ έχω ζητήσει αλλαγές, ε, ξεκινώντας με τα συστατικά ε, το χαρακτηρισμό των οροματικών υλών. Εδώ υποστηρίζω τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν δούμε τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή τη στιγμή, θα δείτε ότι οι κυβερνήσει ανησυχούν γιατί αυξάνει ο αριθμό των ε, τσιγάρων και σχετικών προϊόντων με αρωματικέ ύλε. Η γαλλική κυβέρνηση ήδη έχει απαγορεύσει τέτοια τσιγάρα με γλυκιά γεύση, γιατί φαίνεται ότι προσελκύουν ακόμα και 13 χρόνια, χρόνια. Η κυβέρνηση έχει απαγορεύσει τι περιπτώσει ε, των μεντόλ τσιγάρων και η γερμανική κυβέρνηση ε, ε, επίση έχει τη τσιγάρα μεντόλ. Η, με, τα μεντόλ, η μυνθόλη αν θέλετε, χρησιμοποιείται ευρέω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αν θέλετε να δείτε μετά την δικτύπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε θα καταλάβετε καλύτερα γιατί θέλει να απαγορεύσει τη μυνθόλη η Επιτροπή. Γιατί η μυνθόλη χρησιμοποιείται ακριβώ για να προσελκύσει του νέου το κάπνισμα. Ε, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουμε νέους κινδύνου για την υγεία σε μια έκθεση 100 σελίδων, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μυνθόλη είναι σοβαρή, ε, δημιουργεί σοβαρές παρενέργειες στην υγεία και μεταξύ άλλων ε, ο βήχας κτλ έχουν ε, μελετήσει οι λεκτικές αρχές και η Παγκοσμία Οργάνωση Υγείας ε, αυτά τα φαινόμενα και ιδίως τις συνέπειες που έχει για τους νερούς οργανισμούς ε, η μυνθόλη. Πολύ απλά η μυνθόλη καθιστά το τσιγάρο πιο εύκολο για να το καπνίσει κανεί. Άρα λοιπόν οι επαγγελματίε του κλάδου και οι παγκόσμιε ρυθμιστικέ αρχέ που μελετούν το θέμα λένε ότι γενικότερα τα τσιγάρα με αρωματικέ ύλε θα πρέπει να απαγορευτούν και εγώ το υποστηρίζω. Τώρα σε ό,τι φέρνει την δικαιοθεσία. Η νομοθεσία περί το ε, οι προτάσει της Κομισιόν συγκεκριμένα είναι πολύ καλέ. Όλα τα πολιτικά στοιχεία δείχνουν ότι βοηθούν να αναχαιτήσουμε το φαινόμενο των νέων καπνιστών. Πρέπει όμω να προχωρήσουμε πέρα-πέρα από ό,τι προτείνει η Κομισιόν. Να προσεγγίσουμε μάλλον το σύστημα το Αυστραλιανό ε, και για τα ε, τσιγάρα, τα, στα πακέτα, αλλά και τα στριφτά τσιγάρα. Γιατί το προτείνω αυτό. η τελευταία διαφήμιση που έχουν ως χαρτί στα χέρια τους οι εταιρείε είναι η ίδια ε, η φύρημα που υπογράφει τα τσιγάρα και αυτό θα πρέπει να το απογράψουμε πλέον. Οι εταιρείε καπνού κάνουν και πολύ σκληρά λόμπινγκ στη χώρα μου. Ε, καταχωρίζουν τετρασέλιδες διαφημίσεις στις εφημερίδες ε, γιατί η κυβέρνηση προχωρά αυτή την νομοθεσία αυτή τη στιγμή για την απλή συσκευασία. Τι είναι απλή συσκευασία, θα σας δείξω εγώ τώρα. Κάποιοι συνάδελφοι μου είπαν, βλέπετε αυτή την εικόνα, να την είναι ένα απλό πακέτο. Να, αυστραλιανό απλό πακέτο. Δεν είναι απλό, έχει φωτογραφίες και προειδοποίηση για την υγεία. Να το πακέτο που προτείνει η Κομισιόν, τη συσκευασία προτείνει η Κομισιόν. Ποια είναι η διαφορά είναι η αναφορά στην μάρκα. Στη χώρα μου, η υπηρεσία για τα πρότυπα διαφήμιση ήδη είχε ζητήσει από τι καπνοβιομηχανίε να αποσύρουν κάποιε διαφημίσει γιατί παραπλανούν. Τι λένε στι διαφημίσει του. Μπορούν να κάνουν οποιοδήποτε ισχυρισμού επιθυμούν ότι αυτή η απλή συσκευασία θα οδηγήσει σε αύξηση του, πα, ε, του, του παράνομου εμπορίου τσιγάρων. Όλα όμως λέει ότι παρότι το 50% των τσιγάρων είναι ε, παραποιημένα προϊταπομίσεις γνησίων ε, εταιριών, από την άλλη μεγάλο ποσοστό ε, είναι προϊόντα που μπαίνουν παρανόμως στην νόμιμη αλυσίδα εμπορίου. Και αυτό έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ως αντεπιχείρημα για την αντιμετώπιση ε, για τη μήνυμα αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου α, τσιγάρων. Τα πακέτα απομιμήσεις μπορούν να γίνουν με πάρα πολύ φθηνό τρόπο ήδη. Πώς μπορούν να γίνουν πιο φθηνότερα. Το συνολικό κόστος για ένα τέτοιο πακέτο είναι 15 με 20 ε, λεπτά του ευρώ. Άρα τα προϊόντα απομίμησης και το λαθρεμπόριο τσιγάρων είναι ένα φαινόμενο, ένα πρόβλημα, αλλά δεν είναι αυτό το μείζον. Ουσιαστικά είναι σαν να προσπαθεί να ψάχνει κανείς ψηλοστάχυρα. Νομίζω ότι αν το ρωτήσετε και αυτούς οι κυβερνήσεις θα συμφωνήσουν μαζί μας. Τώρα τα λεπτά, τα slim τσιγάρα θα πρέπει να απαγορευτούν με τη νέα νομοθεσία. Αυτό είναι επίμαχο ζήτημα σε κάποιες χώρες. Γιατί θέλει η Επιτροπή να απαγορεύσει τα τσιγάρα slim αυτά τα λεπτά τσιγάρα, γιατί υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι τα λεπτά τσιγάρα προσελκύουν κυρίω νεαρέ γυναίκε στο κάπνισμα. Αν δεν πιστεύετε εμένα, ακούστε τι λένε οι ίδιε οι εταιρείε. Το 2011 μας λένε η εταιρεία ότι προσπαθούμε δημιουργικά να προσελκύσουμε τον κύκλο των γυναικών χρησιμοποιώντας λεπτότερα ε, και πιο ελκυστικά στη μορφή ε, τσιγάρα. Γι' αυτό χρησιμοποιούνται αυτά τα λεπτά τσιγάρα, τα slim, τα λεγόμενα στις αγορές μας. υπάρχουν διάφορες ε, μάρκες. Εδώ βλέπετε ότι έχουμε ένα πακέτο που μοιάζει και με άρωμα. Ε, ε έχει σχεδιαστεί έτσι, ακριβώς για να προσελκύσει νεαρές κοπέλες. Εδώ βλέπετε άλλο ένα πακέτο μεντόλ που και αυτό ε, είναι πολύ ελκυστικό για τους νέους. Ελπίζω λοιπόν να υποστηρίξετε την πρόταση της Κομισιόν και αυτά που λέω και εγώ και όσους συναδέλφους θέλουμε να παγορεύσουμε αυτά τα προϊόντα στις αγορές μας ώστε να μην χρησιμοποιείται για να δελεάζουν τους νέους ε, στο κάπνισμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού, δεν προτείνω καμιά αλλαγή, συμφωνώ με την Κομισιόν. Διασυνοριακή πώληση προϊόντων καπνού δεν υπάρχει πολύ μεγάλη διασυνοριακή, διασυνοριακό αν θέλετε εμπόριο μέσω ίντερνετ, αλλά πάντως αυτό που υπάρχει δεν είναι νόμιμο. Εννέα κρατημέλη ήδη έχουν απαγορεύσει το διασυνοριακό εμπόριο τσιγάρων και πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι γενικότερο η απαγόρευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, νέα προϊόντα καπνού. Μιλάμε για νέα προϊόντα η Κομισιόν προτείνει σύστημα κοινοποίηση για οποιοδήποτε νέο προϊόν, αλλά επιτρέπει στα κράτη-μέλη να επιλέξουν ε, και την εισαγωγή συστήματος προηγούμενης αδειοδότησης. Ε, στις ε, το FDA έχει τέτοιο σύστημα προηγούμενη αδειοδότησης και δεν επιτρέπει να δοθεί άδεια σε νέα προϊόντα. θα πρέπει να ακολουθήσουμε και εμεί αυτή την προσέγγιση, ώστε να μπορούν οι αρχέ να αναχαιτίζουν την εισαγωγή κακών προϊόντων στην αγορά. Όχι να προσπαθούν να τα βγάλουν από την αγορά όταν υπάρχει ήδη κοινοποίηση ότι υπάρχει πρόβλημα. Φυτικά προϊόντα για τα κάπνισμα. Συμφωνώ και εδώ με την Κομισιόν. Ε, κάτι ξέχασα μόνο να σας πω. Όταν μιλάμε για αρωματικές ύλες στα προϊόντα καπνού, η Επιτροπή απαγορεύει τις αρωματικές ύλες για τα τσιγάρα και τα στριφτά. Δεν αγγίζει όμως τα παραδοσιακά λεγόμενα προϊόντα όπως είναι τα πουρα που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο από ηλικιωμένους. Σας παρακαλώ όμως να σκεφτείτε και το θέμα του ναργιλέα που παραδοσιακά χρησιμοποιούσαν κυρίως πιο ηλικιωμένοι καπνίστες. Όμως βλέπουμε σήμερα και εδώ στα μπαρ στις Βρυξέλλες, στις Εξέλ, κόσμος, νέος κόσμος το χρησιμοποιεί με αργυλέ. Να δούμε κατά το θέμα των αρωματικών ουσιών στον αργυλέ. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Γιατί όταν σου δίνει τον αργυλέ, δεν ε, βλέπεις το πακέτο, όπως όταν αγοράζεις τσιγάρα. Η γαλλική κυβέρνηση και άλλες κυβερνήσεις έχουν εκφράσει ανησυχία για αυτό το φαινόμενο. Θέλω να ακούσω την άποψή σας γι' αυτά. Δεν έχω βάλει ε, τροπολογίες πάντως για το θέμα των ηλεκτρονικών τσιγάρων. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι προϊόντα καπνού. Κάποιοι λένε ότι δεν είναι προϊόντα καπνού. Όχι, είναι προϊόντα καπνού το 90% της νικοτίνης προέρχεται από τον καπνό και συνεχώς αυξάνουν το μερίδιό του στην αγορά. Σε διάφορες χώρες της Ένωσης τη διαφορετική διαφορετικές μεταχείρισης. Κάποιες χώρες απαιτούν έγκριση των ηλεκτρικών τσιγάρων ως φάρμακα, γιατί η νοικοτήνη χρησιμοποιείται εν προκειμένου ως φάρμακο. Αναμφίβολα η νοικοτήνη όμως είναι πολύ εθιστική. Δεν τον φυσφυτεί αυτό κανένας επιστήμων, συλλέγουμε αποδεικτικά στοιχεία για να δούμε τι συμβαίνει με, την, ε, με το τι εκπέμπουν τα τσιγάρα αυτά. Κάποιοι λένε ότι δεν ε, είναι επιβλαβή για την υγεία, όμως αυτό που εκπέμπουν, ο καπνός που εκπέμπουν, ε, ή έχουν, προκαλούν βλάβη στην υγεία. Πάντως οι καπνιστές των ηλεκτρονικών τσιγάρων μπορούν να μειώσουν τη βλάβη σε σχέση με τον, αυτούς που καπνίζουν πραγματικά τσιγάρα. Αυτό πραγματικά υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία προς αυτή την κατεύθυνση. Το πρόβλημα με αυτά τα τσιγάρα πάντως είναι ότι οι τελειωνικά τσιγάρα ε, έχουν πολλές διαφορετικές ποιότητες. Και αφού το εξεταστούν από τι εθνικές αρχέ, έχουν δει ότι κάποιοι δεν περιέχουν καθόλου νοικοτήγνη. Δηλαδή, όταν ελέγχονται, βρίσκονται ελαττωματικά, γιατί δεν υπάρχει καθόλου νοικοτήνη. Λένε, ή δεν λειτουργεί καλά ο μηχανισμό του. Πολλοί αποστέλουν επιστολέ, και εγώ έχω λάβει πολλέ επιστολέ κατά τσιγάρα, και πολλοί με αντιμετωπίζουν εχθρικά εν προκειμένου. Θέλω να πω ότι εγώ δεν θέλω να προωθήσω την απαγόρευση των τσιγάρων. Τα λένε αυτά κάποια λόμπι, δεν ξέρω ποιο τα λέει στον κόσμο. Πάντω εγώ αυτό έχω ακούσει, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν ρυθμίσει για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Το θέμα είναι πώ. Πώ μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα προϊόντα που βγαίνουν στην αγορά είναι ασφαλή, έχουν μια κάποια ποιότητα, ότι οι χρήστε ξέρουν πώ να χρησιμοποιήσουν, διότι αν δεν τα χρησιμοποιήσουν ορθά, αυτοί που τα χρησιμοποιούν για να μειώσουν την βλάβη του καπνίσματο, τελικά θα την καταλήψουν και θα επιστρέψουν στο κάπνισμα. Και θα πρέπει επίση να είναι σαφέ, ότι δεν χρησιμοποιούνται και πάλι, αν θέλετε, για να οδηγήσουν πίσω από την πόρτα ε, νέους και πάλι στο κάπνισμα. Στις 7 Μαΐου θα γίνει ένα εργαστήριο εδώ στο Κοινοβούλιο για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα η ΠΟΗ θα δημοσιεύσει την τελευταία τη μελέτη από το θέμα του απαντά σε τα ερωτήματα πώς είναι οι καπνιστές, τι περιέχει ο καπνός τους, ε, ποιος είναι ο χρήστης, ε, τα στοιχεία για τους νέους ε, σε ό,τι αφορά τη χρήση των τσιγάρων. Λοιπόν, θα περιμένουμε να ακούσουμε και τι έχουν να μα πούν οι ρυθμιστικέ αρχέ από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Φιλανδία που μελετούν πολύ προσεκτικά αυτό το θέμα. Το πώ πρέπει να επιβάλλουμε ρυθμίσει σε ηλεκτρονικά τσιγάρα. Θα ακούσουμε την άποψη των χρηστών Επίσης, είπα ότι δεν έχω υποβάλει ακόμα τροπολογίες γιατί θέλω πρώτα να ακούσω α, α, αυτά που θα υποθούν σε 7 Μαΐου. Γι' αυτό μεταφέρεμε την καταλεκτική μέρα για τις ε, τροπολογίες στις 8 Μαΐου, ώστε και οι συνάδελφοι να μπορούν να ακούσουν αυτές τις μαρτυρίες. Ξέρω ότι ακούτε μαρτυρίες ε, πάντοτε, διαβάζετε ε, αποδεικτικά στοιχεία, είναι καλό να ακούσουμε και αυτές τις μαρτυρίες σε 7 Μαΐου. Είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθήσουμε το θέμα στενά και ορθά. Δεν θέλουμε να επιτρέψουμε ε, να μπουν στην αγορά νέα προϊόντα τα οποία δεν είναι ασφαλή. Γιατί δεν ξέρουμε ακριβώ πώ λειτουργούν. Αυτέ είναι οι αλλαγέ που έχω κάνει, Πρόεδρε. Α, θέλω να ακούσω τι γνώμε του συναδέλφων. Δύο-τρει φορέ έχω δει του σκιώδει σε πολύ επικοδομητικέ συζητήσει. Οι γνωμοδοτήσει των λοιπόν επιτροπών είναι έτοιμε και σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ μαζί μου. Υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία διαφωνούμε και είμαι πολύ καπεπισμένη ότι μπορούμε να βρούμε μια κοινή προσέγγιση για τα θέματα του καπνού. Το ξέρω, όταν μιλώ με του συναδέλφου μου, όλοι συμφωνούν. Θέλουμε να μειώσουμε τον αριθμό των καπνιστών στην Ευρώπη. Σε κάποιε χώρε δυστυχώ η τάση των νέων καπνιστών είναι πολύ ανωδική. Είναι κάτι που πρέπει να σταματήσουμε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μακαβόν. Επτά του μηνό είναι το εργαστήριο αυτό, το workshop. Το έχουμε ανακοινώσει. Σας καλώ όλους να είστε παρόντες. για τα φουγάρα και όχι τα τσιγάρα πλέον, ηλεκτρονικά και άλλα. Και θα ακούσουμε διαφορετικές θέσεις και απόψεις. Είναι ένα θέμα σημαντικό. Πολύ σημαντικό είναι ότι είδου συστατικά μπαίνουν στα τσιγάρα και έχει ιδιαίτερη σημασία να τα δούμε να ενημερωθούμε για την κατάσταση που έχει τώρα μέσα από ένα workshop. Ναι και έχουμε πολλούς ενδιαφερομένους να λάβουν τον λόγο. Θα σας διαβάσω τον κατάλογο. Martin Kellenen, und Martina Andersen und als übrige Redner και άλλους ομιλητές έχω επίσης. Χίπνα, Ντέιβις, Βέστλον, Λίζε, Μπαρτολότσι, Μόκουνάιτε, Morkonaite, Φιέλνα, Κουμπού. Koumoutsantos, äh, Silakakis, Pirillo, Wilmot, Estrella und Rivasi. Habe ich jemanden vergessen? Λυσμόνισα κανέναν. Όχι, καλώς, κλείνει ο κατάλογος. Ο κύριος Καρλ Χάιντς Φλόρενς, σκιώδης από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Μακάβων. Πάντοτε συνεργαζόμαστε πολύ καλά, μας έχει ενημερώσει πολύ καλά δεν έχουμε κανένα παράπονο. Και εύχομαι κάθε επιτυχία. Βεβαίως σε ένα-δυο σημεία δεν συμφωνούμε 100% και θα ήθελα να τα αναφέρω προκαταβολικά, ενώ στα υπόλοιπα ε, στα οποία συμφωνούμε θα είναι πολύ επιγραμματικός. Όσον αφορά την ε, ακρίβεια σε χιλιοστό στην περιγραφή του ε, πακέτου της συσκευασία. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσω. Νομίζω ότι προτιμώ την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν και ακόμα και εκεί πάλι, πάλι σχεδόν μέχρι το χιλιοστόμετρο δίδεται ο ορισμός για το μέγεθος της συσκευασία. Εγώ είμαι, πε, είμαι πεπισμένος υποστηρικτής ε, της ε, ελεύθερης της αγοράς. Δεν νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να υπαγορεύουμε εμείς στην ε, ε, βιομηχανία εάν πρέπει να είναι 8 εκατοστά ύψος ή 10 και 4 ή 5 εκατοστά φαρτο το, το πακέτο των τσιγάρων κτλ. Ή πόσο μεγάλα πρέπει να είναι τα μηνύματα, τα προειδοποιητικά μηνύματα από 50 μέχρι 75%. Ακούμε πολύ διαφορετικές απόψεις στην ομάδα μου, αλλά λέω όχι στο plain packaging και όχι στην πρόταση να πρέπει να ορίζουμε εμείς κάθε λεπτομέρεια. Πρέπει πράγματι να εξηγούμε, να υποδεικνύουμε πώς θα ανοίγει το πακέτο των τσιγάρων. Όταν δίνουμε την ενημέρωση, την πληροφόρηση για τον κίνδυνο του καπνίσματος, εδώ νομίζω ότι είναι το πρόβλημα. Σε αυτό έχουμε ολιγορήσει και εκεί πρέπει να κάνουμε περισσότερη προσπάθεια. Έχω και εγώ τρία παιδιά και ξέρω τι σημαίνει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αφήσουμε τα πακέτα για τα slim. Συμφωνώ με τη Λίντα Μακέβαν. Είναι κάτι το οποίο και λόγω της ελκυστικής εικόνας που δίνει το πακέτο κινδυνεύουν να παρασυρθούν πολλοί νέοι, όπως εκεί και, επίσης και με τα πακέτα αυτά που μπορεί να έχουν ε, τέσσερα ή πέντε τσιγάρα μόνο μέσα και επιπλέον είναι ε, πώς να το πω, γεμισμένα, παραγεμισμένα με διάφορα αρωματικά, διάφορες ουσίες. Σε αυτό συμφωνώ ότι θα πρέπει να απαγορευτούν. για το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Συμφωνώ ότι όντως σε, κάποια, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί κανείς να αγοράσει φερρυπίν ε, στο σταθμό του τρένου τσιγάρα και τότε διερωτώ με γιατί εάν κανείς ε, προτιμάει το ηλεκτρονικό τσιγάρο, γιατί θα πρέπει να τον υποχρεώσω να φτάσει μέχρι το φαρμακείο. Δεν είναι πολύ λογικό αυτό. Ίσως και η καταχώρησή του ως ειδικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει πολύ λογική. Θα πρέπει να το δούμε αυτό λοιπόν. Χαίρομαι επίση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστω και με τρόπο άτολμο επανεφέρει το θέμα των χημικών ουσιών, που, το, δικό μου, το δικό μου μέλημα που χρησιμοποιούνται στα ε, τσιγάρα. Αλλά όπως είπα άτολμα μένα, αλλά έστω είναι μια αρχή και αυτό. Και νομίζω ότι με, τους, ε, με τις λύσεις και τους ορισμούς ε, τις, τους σχετικούς με την ε, γεύση έχουμε βρει μια λύση για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ενεργείας των δικηγόρων γιατί φαντάζεστε τι δουλειά θα σημαίνει το να ερμηνεύσει κανείς την μία ή την άλλη γεύση και τον τρόπο με τον οποίο η χημική βιομηχανία μπορεί να διαμορφώσει το τελικό αισθητήριο, την τελική αίσθηση μάλλον που θα δίνει στο στόμα ένα, ένα συγκεκριμένο υλικό, μια συγκεκριμένη ουσία θα υπάρχουν πολλά προβλήματα προς την Ερμηνεία. Εγώ θα προτιμούσα να είναι πολύ πιο συγκεκριμένη η αναφορά σε μια ουσία που θα απαγορεύεται και από εκεί και πέρα να μην κοιτάμε τι είδους τελικό αποτέλεσμα και τι αίσθηση δίνει. Ένας κατάλογος χημικών επικίνδυνων χημικών ουσιών είναι πολύ πιο ασφαλής λύση για μένα. Είναι σύστημα που ισχύει σε κάποια κρατημέλη ήδη και δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να το υποτιμούμε. Για τα slim μίλησα ήδη, ε, προειδοποιητικά μηνύματα, ως προς τα ποσοστά δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ, αλλά εν πάση περιπτώσει μια διαδικασία είναι αυτό για τον ε, καπνό για μάσημα ε, είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό τοπικό προϊόν. Έχουμε φερειπίν στην Νότια Γερμανία τον ε, καπνό για, για τη μύτη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι βγαίνει αυτή η αναφορά. Νομίζω ότι πάνω από 40 με 50% του παράνομου ε, μπορείου τσιγάρου περνάει από νόμιμα παραγόμενα τσιγάρα της ε, Εάν δεν ε, πληρείται η ποσόστοση την οποία θέλουν για να πάρουν την ενίσχυση, τότε αυξάνουν στα, τα νούμερα στα χαρτιά, παίρνουν την ενίσχυση και τα υπόλοιπα τσιγάρο περισσεύουν, πάνε ως παράνομο, ως λάθρεμπόριο στα ε, κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Το μέγεθος του ε, πακέτου της συσκευασία είναι προτιμότερη πρόταση Επιτροπής. Για τα ποσοστά μπορούμε να συζητήσουμε και θα συζητήσουμε. Συμφωνώ να υπάρχουν γραπτές προειδοποιήσεις και ενδεχομένω και με αναφορά μιας ειδική γραμμής τηλεφώνου. Μου φαίνεται λίγο ε, υπερβολικό το να θέλει κανείς να ελέγξει το πόσο μεγάλη θα είναι η διαφήμιση του παραγωγού μια συγκεκριμένη ε, επιχείρηση. Αυτό νομίζω δεν χρειάζεται νομοθέτημα για να το ελέγξει κανείς. Στη τελευταία ανάλυση αυτά μπορούν να καταγραφούν μέσα από τον συλλογισμό της εταιρείας πολύ ξεκάθαρα, πόσο ποσοστό δηλαδή δίνει στην ε, ε, διαφήμιση και ως εκ τούτου να γίνει ο έλεγχος. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε και στη συνεργασία με τη συνάδελφο βεβαίως, αλλά πάνω πολλά και με το Συμβούλιο, να καταλήξουμε σε μια καλή λύση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Καρν Χάιντς Φλόρεντς. Μάλιστα. Επόμενος ομιλητής, εκ μέρους της ομάδας Άλντε, η Φρέντερικ Γκρίς. Merci beaucoup. ευχαριστώ πολύ και εγώ θα είμαι πολύ σύντομη. Συντομή, θα ευχαριστώ τη Λίντα για την πολύ καλή δουλειά της και για την πολύ καλή συνεργασία μεταξύ τη ηγητρίας και των σκιωδών. Με πολύ ενδιαφέρον ε, παρακολούθησα, διάβασα την ε, εκθεσή της. Καμιά από τις 56 τροπολογίε τη, δεν υπολείπεται φιλοδοξία σε σχέση με αυτές, με τις ε, προτάσεις δηλαδή, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γι' αυτό την ευχαριστώ για την πολιτική στάση της. Ε, θα περιοριστώ στην, στα ουσιαστικά στοιχεία γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Στο άρθρο 6 βεβαίως για τα, για τα συστατικά συμφωνούμε με την ενίσχυση των ε, διατάξεων για τα είδη καπνού που καταλαβαίνουν περισσότερο οι νέοι, κατά προτεραιότητα, 24-29 τροπολογίες συγκεκριμένα. Επίσης και η Λίντα τον ανέφερε, είμαστε υπέρ της ε, προηγούμενης αδειοδότησης των προϊόντων καπνού 48 έως 51 τροπολογίες για το άρθρο 17. Ανέφερε η Λίντα ήδη τις ε, θέσεις των ΗΠΑ και της FDA. Επίσης ε, η υγειονομική διάσταση, labeling, συσκευασία. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι είναι φιλόδοξη η πρόταση Επιτροπής γιατί αυτή την υποχρέωση να συνδυαστεί η προειδοποίηση με τη φωτογραφία την επεκτείνει στα 27 κράτη-μέλη, πράγμα το οποίο δεν αντιστοιχεί στις παραδόσεις, πάνω σε 75% του ποσοστού επί της συσκευασίας. Ε, θα θυμάστε πόσο, πόσο νερό έχει κυλήσει από τότε που ξεκίνησε αυτή η πρώτη προσπάθεια με την πρώτη οδηγία. Για να επανέλθω στο ε, στο θέμα που είπα θα πρέπει να κοιτάξουμε τα ποσοστά μπρος, πίσω, ε, ποσοστό επί της συσκευασίας κτλ. Είναι η συζήτηση που κάναμε πριν από 10 χρόνια και θα σας θυμίσω ότι είχαμε δει ήδη από κάποια πρωτότυπα συσκευασία που κυκλοφορούσαν στην καπνοβιομηχανία είχε γίνει ήδη συζήτηση ακόμα και για το μελάνι ή για το, το πλαίσιο ε, και κάποιε λέγανε είμαστε τρελοί. Ε, είδαμε λοιπόν τα πρότυπα της ε, ε, καπνοβιομηχανίας που κυκλοφορούσαν γιατί μπορεί Εμεί να μην είμαστε ικανοί να κάνουμε αυτή την ε, εικονική απάτη, την ο, ο, οφθαλμαπάτη, αλλά η καπνοβιομηχανία κατάφερε να κάνει μια πολύ εντυπωσιακή οφθαλμαπάτη, βάζοντα είτε φιλιγκράν, είτε θαμπά, είτε διάφορα άλλα ε, στοιχεία πάνω στη φωτογραφία και στην διαμόρφωση της συσκευασία που ε, τελικά αλλίωναν το μήνυμα και τις ε, ε το, το επιδιωκόμενο μήνυμα. Ε, συμφωνώ με την κυρία Μακάβαν λοιπόν στα περισσότερα, αλλά θα ήθελα να πω το εξή, γιατί θα μετατραπώ σε συνήγορο του ε, διαβόλου τώρα. Ε, στο θέμα αυτό, γιατί δεν αφήνουμε στα χέρια των κρατών μελών για το υπόλοιπο 25%. Στα 25 κρατημέλη υπάρχουν πολλές φορές ακόμη μόνο προειδοποίησεις και δεν υπάρχουν φωτογραφίες. Τώρα μιλάμε για υποχρεωτική κάλυψη μαζί με, το, με φωτογραφία του 75% αλλά το 25% γιατί δεν μπορεί το κράτος να κάνει κάτι επιπλέον. Τώρα για τον λεγόμενο Ναργιλέ. Είναι πολύ ε, βλαπτική για την υγεία με πολύ υψηλότερο ποσοστό μονοξυδίου του άνθρακα από ό,τι στα λοιπά προϊόντα καπνού είναι αυτό του, της εξάτμισης του αυτοκινήτου, η ποιότητα του μονοξυδίου. Άρα έχω τροπολογίες 6 και 10 που έχουν στόχο να είμαστε ακόμη πιο αυστηροί. Προσπαθώ πολύ γρήγορα να τα κάνω. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα τώρα. Θα συμφωνήσω με τη Λίντα και τον Καρλ Χάιντς Περιμένω να δούμε το workshop, το εργαστήριο που έχουμε σε έξι του μηνό. Δεν έχει οριμάσει η συζήτηση. Καταρχά, εγώ μόνη μου δεν έχω κατασταλάξει, αλλά και στην ομάδα των φιλελευθερών επίση. Ε, ή θα είναι η ιδέα τη ε, αποκοπή τη ε, απεξάρτησης, είτε θα είναι η ιδέα της υποκατάστασης, κάπως πρέπει να συστήσουμε το θέμα αυτό του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Το άρθρο 18 πάντως είναι πολύ ακριβό, είναι μία τάση να χαρακτηρίζεται ως ε, καταστροφική ή ως υπέτειο για τα πάντα, ενώ είναι μία λύση που θα μπορούσε κάποιος να τους βοηθήσει να εγκαταλείψουν το κάπνισμα. Καταρχάς λοιπόν, εάν είναι ποσοστό, το ποσοστό νοικοτήνης ισοδύναμο με αυτό που βλέπουμε σε άλλα ε, προϊόντα απεξάρτησης, όπως τα πάτσου της νοικοτήνης, γιατί όχι. 8 με 10 μιλιγκράμμ, ε, δεν ξέρω εάν ε, μπορώ να δεχθώ τις Επιτροπής και αυτοί οι ατμοκαπνιστές, θα λέγαμε, vapoters στη Γαλλία, ε, εν πάση περιπτώσει μπορούν να διαλέξουν μια λύση που δεν έχει τόσο μεγάλο ποσοστό νικοτίνης και με πολύ μεγάλη προσοχή θα κοιτάξουμε την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων αυτών που δεν έχει εξεταστεί ακόμη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρίς. Κάρλ Σλίτερ, τώρα εκ μέρους των Πρασίνων. Eh, Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για την πρότασή του. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την πρόταση αυτή, ιδιαίτερα για ότι έχει σχέση με τι θα αναγράφεται πάνω στο πακέτο. Και πραγματικά ελπίζω αυτό να διευρυνθεί σε όλες τις μορφές καπνού, όχι μόνο στα τσιγάρα και τα στριφτά. Αν δούμε τους ε, λόγους, τις αιτίε πίσω από όλα αυτά τότε θα δούμε ότι προσπαθούμε να αποτρέψουμε τα παιδιά και τους εφήβους από το να αρχίσουν το κάπνισμα και σε κάποιο βαθμό να βοηθήσουμε εκείνους που ήδη έχουν αρχίσει το κάπνισμα να μην στρατολογούν άλλους. Δεν θέλουμε νέα γενιά καπνιστών. Δεν αντέχουμε οικονομικά μια καινούργια γενιά καπνιστών. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εάν εφαρμοστεί τότε, θα έχουμε καθαρά κέρδη. Πραγματικά, θα έχουμε φορολογικά έσοδα. Και όχι όπως λένε απώλειες. Μας λένε ότι άμα απαγορεύσουμε το κάπνισμα και μειωθεί ο ρυθμός των καπνιστών θα έχουμε λιγότερα, λιγότερα έσοδα. Όχι όμως. Αυτοί οι καπνιστές θα κατευθυνθούν αλλού, θα χωράσουν άλλα προϊόντα. Το θέμα όμως δεν είναι το οικονομικό κέρδος, είναι το κέρδος της υγείας. Το περισσότερο κομμάτι από την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται σε νούμερα. Εγώ πιστεύω ότι το κέρδος μπορεί να είναι πάνω από 25 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο με αυτά τα μέτρα κατά του καπνίσματος. Δεν θέλω να ληφθούν μέτρα για τον καπνό, αλλά ας ανεβάσουμε τη φορολογία. Όχι, αυτό είναι παράλογο. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως πρέπει να πάμε ακόμα παραπέρα από αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πολύ καλή πρόταση η πρόταση της Κομισιόν και η πρόταση της Λίντα είναι πάρα πολύ καλή, αλλά θέλω να σας πω κάτι για αυτό το τυποποιημένο πακέτο. Το έχω μπροστά μου. Από... Αυτό είναι ένα τυποποιημένο πακέτο από τη Σουηδία, η οποία δεν είναι και η πρώτη στον έλεγχο αυτή τη στιγμή των ε, καπνών. Αυτό εδώ είναι ένα παράδειγμα ε, καπνού χωρίς πρόσθετα συστατικά. Σε ένα φυσικού χρώματος καφέ πακέτο. Εδώ είναι ένα βέλγικο πακέτο, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε γυναίκες. Αυτό το μικρό δηλαδή, το ροζ. Και ξεκάθαρα, το ροζ πακέτο απευθύνεται στις γυναίκες. Είναι προφανές. Και έχουμε και ακόμα περισσότερες ενδείξεις οι οποίες μας μαρτυρούν ότι η καπνοβιομηχανία κατευθύνεται και στοχεύει τις γυναίκες με ωραία προς, ε, χρώματα, με λεπτά σχήματα, με γεύσεις. Καρλ Χάινς, συμφωνώ και εγώ το απεχθάνομαι όταν ρυθμίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα πάντα μέχρι τη τελευταία στρανίδα. Όμω πραγματικά η καπνοβιομηχανία εδώ πέρα έχει πολύ περισσότερου εμπειρογνώμονε από ό,τι έχουμε εμεί. Του πληρώνει για να δουλεύουν ολική απασχό... Ε, ε, για να δουλεύουν full time για να βρίσκουν τα παραμικρά κενά και να τα διορθώνουν. Γι' αυτό λοιπόν πραγματικά πιστεύω φτάνει. Πρέπει εδώ να μην αφήσουμε κανένα παραθυράκι ανοιχτό, να τα κλείσουμε όλα, μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να μην έχουν, όπως είπες και εσύ, δουλειά οι δικηγόροι μετά. Για να μην μπορεί η καπνοβιομηχανία να κάνει διαφημίσει σε παιδιά. Ξέρετε ότι το 60% των καπνιστών αρχίζουν το κάπνισμα πριν τα 18. Δεν είναι δική τους επιλογή ενσυνείδητη λοιπόν. Εμείς οι ενήλικες που αποτελούμε τους ε, ε, απασχολούμενους στην καπνοβιομηχανία, που ευθυνόμαστε για τον εθισμό των παιδιών αυτών, πρέπει πραγματικά να φροντίσουμε να μπει ένα τέλος. Και η Λίντα μίλησε για τους ναργιλέδες. Παλιά ε, ναργιλέδες κάπνιζαν μόνο οι παππούδες, τώρα έχει γίνει μόδα. Μόδα στους νέους, ανάμεσα στους νέους. Είναι νέα, νέο, νέα πόρτα που θα τους βάλει στο κάπνισμα. Το ίδιο και με τα σλίντσιγάρα. τσιγάρα και τα τσιγάρα μενθόλης. Κάνει το κάπνισμα πιο εύκολο σε κάποιον που δεν το έχει συνηθίσει. Δηλαδή καταστέλει αυτήν την, την αντίδραση, τη φυσική αντίδραση του, του σώματος να πνίγεται. Και τον διευκολύνει λοιπόν να αρχίσει το κάπνισμα. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Δεν μπορούμε να, επιστρέψουμε, να, να επιτρέψουμε πρόσθετα τα οποία θα κάνουν το κάπνισμα πιο εύκολο παρομοίως και με το διαδικτυακό εμπόριο από το ίντερνετ. Πρέπει να το απαγορεύσουμε πλήρως, όχι μόνο το διασυνοριακό, το εμπόριο στο ίντερνετ γενικότερα. Και υπάρχουν ορισμένα επιχειρήματα τα οποία τα θεωρώ μη ευσταθή για το λαθρεμπόριο Όσον αφορά το λαθρεμπόριο πρέπει να δούμε και την πλευρά της προσφοράς και την πλευρά της ζήτησης, να τις δούμε και τις δύο. Η Κομισιόν έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες για την ασφάλεια, για να αποφευθεί το λαθρεμπόριο. Εμείς πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα παραπά, πέρα από αυτά που προτείνει η Κομισιόν. Αυτό το τυποποιημένο πακέτο με τις λεπτομέρειες είναι πολύ πιο δύσκολο να παραποιηθεί από ότι τα πακέτα που υπάρχουν σήμερα και αυτό είναι το αντίθετο από ό,τι υποστηρίζει η Κομισιόν. Επίσης, παρομοίως για τις χώρες οι οποίες έχουν πιο αυστηρούς ελέγχους στα σύνορά τους, οι οποίες με ε, μείωση του λαθρεμπορίου θα έχουν μεγαλύτερα έσοδα από τις πωλήσει τσιγάρων. Τώρα όσον αφορά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Σήμερα τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ρυθμίζονται από πάρα πολλούς διαφορετικούς φορείς και αυτό είναι το πρόβλημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν κάποιος καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο, ρουφά και το υγρό που έχει μέσα και κινδυνεύει να πάρει υπερβολική δόση νοικοτήνης και άλλων τοξικών ουσιών. σε πολύ μικρές ε, ποσότητες κάποιες από αυτές ε, τις ουσίες επιτρέπονται, όμως όχι στην ποσότητα που περιέχεται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Αυτές οι ποσο... Αυτά τα συστατικά περιέχονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν προορίζονται για εισπνοή και έχουν τελείως διαφορετικά αποτελέσματα λοιπόν στον ανθρώπινο οργανισμό από ότι με την ε, εάν ληφθούν Τώρα, το να θεωρηθούν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ε, φαρμακευτικό, παραφαρμακευτικό προϊόν με βρίσκει διάφωνο. Χρειαζόμαστε βέβαια σε κάθε περίπτωση μία μεταβατική περίοδο, μία μεταβατική περίοδο αρκετών ετών, με αρκετό χρόνο έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε τις λεπτομέρειες. Τώρα, Σουηδία. Η Σουηδία έχει ένα μεγάλο θέμα με τον καπνό που λαμβάνεται στο στόμα, από το στόμα. Το θέμα λοιπόν ε, του καπνού σνούς ε, είναι μεγάλο θέμα για τους Σουηδού και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σχέση Σουηδία και Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τότε που μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή ε, μάλιστα Σουηδία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την προϋπόθεση να μην υπάρχει απαγόρευση αυτού του καπνού σνούς. Θα έχουμε λοιπόν δι πρόβλημα δημοκρατίας να απαγορευτεί αυτό ο καπνο. Η Σουηδία είπε ναι μόνο και μόνο υπό αυτή την προπόθεση. Και τώρα τι, Τώρα δηλαδή, εάν πούνε στους Σουηδούς όχι, σας είπαμε ψέματα, θα έχουμε θέμα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια λύση, έστω μια λύση μόνο για τη Σουηδία. Έστω να αναλάβει μόνο, μόνο της, η Σουηδία την ευθύνη για αυτόν τον καπνό. Σήμερα υπάρχει αυτός ο καπνός με πάρα πολλές ε, διαφορετικές γεύσεις. Με φρούτα, με μούρα, με ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Και εντάξει, ορισμένοι ισχυρίζονται ότι ο καπνός νους είναι λιγότερο επικίνδυνο. Δεν πάβει όμως να είναι, να είναι επικίνδυνο, δεν είναι τελείως ακίνδυνος. πραγματικά στην περίπτωση της Σουηδίας πρέπει να βρούμε μια καλή συμβιβαστική λύση και όχι απαγορεύσεις. Είναι σαφές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σλούτσερ. Κάνουν Ευχαριστώ πρόεδρε. Αισθάνομαι ανεπαρκή στη συζήτηση αυτή. Δεν έχω πολλές φωτογραφίες και κοριτσίστικα πακέτα τσιγάρου να σας δείξω. Ζητώ συγγνώμη που είμαι τόσο στεγνός, αλλά ε, τα εποπτικά μέσα τα αφήνω στον, ε, στην ε, Λίντα και τον Κάρλ. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, με πολύ ενθουσιασμό. Ομάδες εργασίες, εργασίας, ε, ε συμμετοχή στα διάφορα εργαστήρια των ε, παραγόντων της αγοράς κτλ. Και ευχαριστώ πολύ για τα διάφορα θέματα με τη σειρά. Συστατικά. Συμφωνεί η ομάδα μου με την Επιτροπή και τη Λίντα ότι κατευθυντήρια ο στόχος θα πρέπει να είναι να μην αρχίζει να καπνίζουν. αυτό πρέπει να αποτρέψουν. Όπως είπε και ο Επίτροπος, ο καπνός πρέπει να είναι σαν καπνός ε, και να έχει γεύση καπνού. Να μην έχει γεύση ούτε βανίλιας ούτε κάποιου ε, καραμέλα σαχαρωτού για να απευθύνεται στον ε, έφηβο και τον νέο. Αυτό πρέπει νομίζω να το προσδιορίσουμε ίσω και με απαγορευτικές διτάξεις. Πάντως πρέπει να επαγρυπνούμε ώστε οι προτινόμενη απαγόρευση ενδεχομένως διαθέσει στην αγορά θα είναι σύμφωνη με την ανθεωρημένη οδηγία και θέλω να ακούσω τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ορισμένα ζητήματα στην, ε, που ενδεχομένω υπάρχουν στην ε, υλοποίηση, στην εφαρμογή δηλαδή. Λυπούμε που δεν θέλει να περιορίσει τα ουσιώδη ε, εθιστικά η η συγγητρία αφήνει τα διάφορα σιγαρέτα, ε, τσιγα, ε, πουρα, πουράκια κλπ. Ε, είδη καπνού εκτός του πεδίου εφαρμογής. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι απευθύνεται, απευθύνονται αυτά τα πουρα και πουράκια σε ένα πιο ηλικιωμένο κοινό και λιγότερο στους νέους. Η ομάδα μου υποστηρίζει την ιδέα της ενίσχυσης των προειδοποιήσεων για την υγεία, ε, με φωτογραφίες, με 75% κάλυψη στη συσκευασία και για τον καπνό για τύλιγμα. Εάν χρειάζεται θα πρέπει να δίνετε δυνατότητα στα κράτη-μέλη να είναι πιο αυστηρά. Αυτό άλλωστε υπαγορεύει και η επικουρικότητα. Τέτοια μέτρα μπορούν και έχει αποδειχθεί ότι μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Οι και οι Καναδά είναι τα παραδείγματα. Επίση, Αντιλαμβάνομαι ποιες είναι οι προθέσεις της συγκεντρίας, αλλά εκεί όπου ζητεί η υποχρεωτική ε, με βάση προδιαγραφές τυποποιημένη συσκευασία στο πρότυπο των ε, Αυστραλών, νομίζω ότι ξεπερνάει το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας. Εδώ έχει νομική βάση την εσωτερική αγορά και άρα κάθε είδου τυποποίηση υποχρεωτική θα πρέπει να απαγορεύεται ή να αποκλείεται στην περίπτωση αυτή. Ούτε ελάχιστο ρυθμό σιγαρέτων ή μεγέθου ε, εκατοστών δηλαδή μπορούμε να υπαγορεύσουμε. Άλλωστε ούτε η αναγκαινότητα ούτε η αναλογικότητα μπορούν να αποκλειεται στην περιπτωση αυτη ουτε ελαχιστο ρυθμο σιγαρετων η μεγεθου εκατοστων δηλαδη μπορουμε να υπαγορευσουμε αλλωστε ουτε η αναγκαιροτητα ουτε η αναλογικοτητα μπορουν να υπαγορευουν μια τέτοια επιλογή. Στο ελαφρεμπόριο. Ξέρουμε ποιε είναι οι δυσκολίε. Με ό,τι και να λέμε μπορεί να διωγγωθεί το φαινόμενο αυτό. Εγώ επισκέφτηκα λιανοπολιτή της περιοχής μου ε, πριν από λίγο καιρό για να συστήσουμε τα προβλήματά τους. Ε, ο άνθρωπος βγήκε στον δρόμο λοιπόν και μου γύρισε με μια σειρά από πακέτα σιγαρέτων με κυριλική γραφή, δεν ξέρω από πού τα βρήκε, έτσι με ωραία κίτρινα λαμπερά χρώματα. Ο καπνό ε, γιατί λίγο από ό,τι φαίνεται, ο περισσότερο είναι λαθρέο. Από άλλε χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή είναι πολύ ψηλή φορολογία στον Ηνωμένο Βασίλειο, έρχεται ε, από τι άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εκτό. Και βέβαια πολλέ φορέ έχουμε τελείω ε, πλαστά προϊόντα, απομίμηση δηλαδή προϊόντα, τα οποία μπορεί να είναι και φλαβερά για την υγεία. Αλλά πάντω είναι πολύ φθηνά. Αυτά πρέπει να τα αναλογιστούμε λοιπόν. Πρέπει να αναλογιστούμε λέει, τι συνέπειες των όσων προτείνουμε και θα ήθελα επί τη ευκαιρία να παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί για το πώς θα πρέπει να χειριστούμε το θέμα των τρίτων χωρών, το ζήτημα της ε, σήμανσης και της συσκευασία πιστεύω ότι είναι αντίθετο ε, στις αρχές του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και μπορεί να καταδικαστεί ως ε, μη δασμολογικός φραγμός. Επίσης, θα πρέπει ό,τι μέτρα συχθούν να εξασφαλίζουν την ασφάλεια δικαίου ε, χρειάζεται επι, επαλήθευση, χρειάζεται έλεγχος, χρειάζεται ενημέρωση του λιανοπολιτή και η απαγόρευση ορισμένων πωλήσεων δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι σύμφωνη με τους στόχους για τα καινούρια προϊόντα καπνού. Ε, novel tobacco products. Ναι, θα πρέπει να βεβαιωνόμαστε, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι πληρούν τις προδιαγραφές της και συμμορφώνονται στις αρχές της οδηγίας. Εάν δεν γίνεται αυτό, ενδεχομένως και να χρειαστεί να εισαγάγουν τα κράτη-μέλη κατά περίπτωση ε, οι προϋποθέσεις προηγούμενης αδειοδότησης, εφόσον υπάρχουν ανησυχίες και για την ε, επικουρικότητα μπορεί κάθε κράτο να κάνει διαφορετικέ ρυθμίσει και ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δεν είναι υποχρεωτική η προκαταρκτική ε, αδειοδότηση δυνάμει τη προτάσεώ του. Ε, για το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Το ακανθόδησε αυτό το θέμα, το παρακολούθησα πολύ στενά. Παρακολούθησα και το πρώτο σεμινάριο που είχε οργανώσει η συγγήτρια και είδαμε μία σειρά από ανησυχίε των Ε, ψηφοφόρων της εκλογικής μου περιφέρειας. Δεν είναι πιστικό το ότι είναι ε, φαρμακευτικά προϊόντα και ότι θα πρέπει από αυτή την οδηγία το, για τα φαρμακευτικά δηλαδή να υπάρχουν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Νομίζω ότι η ουσία είναι εάν μπορεί να αποτελέσει αυτό ένα ε, μέσο να αρχίσει κανείς το κάπνισμα, ένα μέσο να προσελκυθεί δηλαδή ένας νέος καπνιστής, ή όχι. Εγώ νομίζω ότι ισχύει το αντίθετο, δηλαδή είναι υποκατάστατα, μπορεί να φέρουν αποτέλεσμα, να βοηθήσουν κάποιον ε, να σταματήσει, να κόψει το κάπνισμα. Πολλοί ήταν οι ψηφοφόροι και νομίζω ότι ήταν ειλικρινεί που μου έγραψαν για να πούν ότι κινδυνεύουν να ξαναγυρίσουν στο κάπνισμα εάν δεν έχουν ευκαιρή πρόσβαση στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Πρόκειται για μια αγορά η οποία έχει ξεκινήσει αρρύθμιστη αυτή τη στιγμή. Ναι, ευχαριστώ Κάρλ. Ναι, είσαι να μου κοπανίσει το σφυράκι, ξέρω. Ε, δεν υπάρχουν επιχειρήματα λοιπόν που να δίνουν αποτελεσματικά καταληκτικά συμπεράσματα για το πώς είναι αυτοί που βοηθήθηκαν και να σταματήσουν οι άλλες συνέπειες στην υγεία του ανθρώπου. Είναι μάλλον εμπειρική η καταγραφή κάποιων συνεπειών. Ως εκ τούτου δεν θεωρώ ότι η οδηγία για τα φαρμακευτικά προϊόντα είναι το κατάλληλο πεδίο για να ρυθμίσει το θέμα αυτό. Η ασφάλεια προϊόντων και άλλα, ε, άλλα νομοθετήματα για ε, δηλητήρια κτλ. μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμες βάσεις. Ίσως να αποδειχθεί ότι είναι πολύ δύσκολη, επειδή είναι πολύ η μικρή παραγωγή που παρασκευάζουν τα ηλεκτρονικά αυτά τσιγάρα, να φανεί πολύ δύσκολη η ρύθμιση του συνομοθετική, χωρίς να περιμένουμε και, ε, να, και να δούμε ενδεχομένω αναπάντεχες ή και αντίξωες συνέπειες. Κοινοποίηση, ενημέρωση, προφανώς ε, προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Για το Σνούς θα είχα να πω δύο λόγια, αλλά και ο Κρίστοφερ περιμένει. Θα τα καλύψει φαντάζομαι. Αντιλαμβάνομαι ποια είναι τα δικά του μελήματα, αλλά θα τα αφήσουμε. Ο κύριος Άντερσεν, η κυρία Άντερσεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να σε ευχαριστήσω και εγώ. Ευχαριστώ την για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ήδη οι πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πολύ φιλόδοξη. Τώρα γίνεται ακόμη πιο φιλόδοξη με τι προτάσει τη συγκεντριά. Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ακόμα πιο φιλόδοξοι και να ζητήσουμε πάνω το 95% κάλυψη ε, του πακέτου με προειδοποίησει για την υγεία. Να ζητήσουμε το 80% του πακέτου. Γιατί όσο πιο μεγάλη είναι η προειδοποίηση, τόσο μεγαλύτερε οι συνέπειε, οι επιπτώσει. Ας είμαστε πιο φιλόδοξοι. Η απόφαση για τροποποίηση τη οδηγία για να έχουμε πλήρως τυποποίηση της συσκευασία σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΗ και τις κατευθυντήριε γραμμές της νέας σύμβασης πλαισίου για τον έλεγχο του καπνού είναι η σωστή προσέγγιση. Και η τελευταία φάση στην οποία μπορούσαν να, να κάνουν διαφήμιση οι είχαν σκοπό να προσελκύσουν ε, τα νεότερα άτομα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί και περιοριστικοί. Ήδη ιστορικά έγγραφα τη βιομηχανία δείχνουν ότι έχουν ε, καταβάλει τεράστιες προσπάθειες και έχουν χρησιμοποιήσει ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για να κάνουν αυτή τη διαφήμιση. Ο ισχυρισμό τη βιομηχανία, ότι δεν ενδιαφέρεται να προσελκύσει νέους, νεαρούς καπνιστές, αλλά ότι θέλει μόνο να αλλάξει τη μορφή ε, και την εικόνα που δίνει η, η, η φίρμα τους, η μάρκα τους, ε, είναι κάτι που δεν μπορούμε να πιστέψουμε. Το συζητήσαμε και σήμερα και σε προηγούμενες συναντήσεις, το έχουμε δει και στα ιστορικά έγγραφα από τη βιομηχανία. Για αυτούς τους λόγους θέλουμε και εμείς τροπολογίες που να προβλέπουν απαγόρευση από της διαφήμισης των προϊόντων στα σημεία πώληση. Ήδη το ξεκινήσαμε αυτό στην Ιρλανδία το 2009 και ήδη βλέπουμε τα ωφέλη ε, καθώς μειώνεται το ποσοστό ε, καπνιστών μεταξύ των νέων. Ένα άλλο επιμαχρό ζήτημα ε, χαρακτηριστικών ε, αρωματικών ουσιών. Θέλουμε να πάμε παραπέρα από αυτή την πρόταση της Κομισιόν. Πρόκειται για ουσίες που βοηθούν ε, τα προϊόντα καπνού να γίνουν πιο ελκυστικά για τον ουρανίσκο. Μια πλήρης απαγόρευση αρωματικών υλών θα ήταν κατάλληλη. Και όχι μόνο αυτό που προτείνει η Επιτροπή. Όπως προτείνει η Κομισιόν στην οδηγία αναφέρει ότι ε, η πρόσθετη ουσία είναι μία ουσία που θα πρέπει να αναφέρεται στα συστατικά, στο συσκευαστικό του πακέτου εκτός από τα φύλλα ε, του ε, καπνού. Με αυτόν τον ορισμό και η ζάχαρη είναι πρόσθετη ουσία. Μια ουσία που καθιστά πιο ελκυστικό το προϊόν στον ουρανίσκο. Ακόμα και αν δεν είναι σαφής ποια είναι η γεύση του ίδιου του προϊόντος, γίνεται πάντα προσπάθεια, ακόμα και ο ανώθευτος καπνός, να γίνει πιο ελκυστικός γευστικά. Θα πρέπει λοιπόν οι πρόσθετες ουσίες να πούν σε ένα συγκεκριμένο κατάλογο και να πούμε ποιε είναι αυτέ τι πρόσθετε ουσίε που είναι απαραίτητε για την Παρασκευή. Έπειτα, πρόσθετε που είναι τοξικέ ή που βοηθούν τον πιο περισσότερο εθισμό θα πρέπει να απαγορευτούν. Τέλος, και εγώ είμαι τη γνώμη ότι η νομοθεσία για την τοποθεσία θα πρέπει να διευρυνθεί και στα πουρα και στα σιγαρέτα και τις πίπες. Το να σταματήσει κανεί το κάπνισμα οποιαδήποτε στιγμή στη ζωή του σίγουρα θα του δώσει ωφέλη για την υγεία. Και ιδίω αυτό αφορά του νέου θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και την περίπτωση των ηλικιωμένων καπνιστών. Θα περιμένω την ακρόαση της 7ης Μαΐου για να συζητήσουμε και με τους συναδέλφους τι διδάγματα μπορούμε να αντιλήσουμε σε αυτή τη φάση, πάντως ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, μετά από τις πολλές συζητήσεις και το ε, υλικό που έχουμε στη θέση μας επί του θέματος, πείθουμε όλο και περισσότερο ότι αυτά τα προϊόντα δεν μπορούν να εξαιρεθούν από μια πιο αυστηρή νομοθεσία. Σε αυτή τη φάση λοιπόν ευχαριστώ και πάλι την εισηγήτρια και την ομάδα της για τη δουλειά που έκανε και ιδίω τον τρόπο με τον οποίο έχει προσεγγίσει τους κοιόδης. Θεωρούμε ότι η βιομηχανία και όλοι ε, έχουν την ευκαιρία να πούν ε, την άποψή τους ε, και σε αυτή την ακρόαση. Θερμά συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Πάντα κάθομαι σε αυτήν εδώ την καρέκλα του Προέδρου και έχω πολλούς ομιλητές και λίγο χρόνο να τους δώσω. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ τη συνεργασία σας. Δείξτε κατανόηση προς τους συναδέλφους σου. Δυστυχώς μόνο ένα μισή λεπτό θα έχει ο καθένας. Ξέρω ότι έχετε να πείτε πολλά περισσότερα, όμως έχουμε τόσους πολλούς έτσι ώστε αν μιλήσετε όλοι το χρόνο που θέλετε δεν θα μπορείτε η Κομισιόν της Υγήτρια να απαντήσει. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εγώ θα τηρήσω το 1,5 λεπτό. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι εδώ μιλάμε για ένα θέμα υγεία. Και οι καπνιστέ πρέπει να σταματήσουν να καπνίζουν και οι νέοι να μην αρχίσουν το κάπνισμα. Αλλά δεν πρέπει όλα να τα βλέπουμε, αν θέλετε, να τα βάζουμε σε δύο τσουβάλι. Το θέμα δεν είναι το μέγεθο που θα πρέπει να έχει το τσιγάρο. Το θέμα είναι ο καπνό, και καπνό καπνού, τα συστατικά του τσιγάρου και θα... η ενημέρωση των νέων. Ε, η πληροφόρησή τους ε, στα σχολεία. Το να πεις ότι ένα κοριτσάκι θα αρχίσει να καπνίσει γιατί είναι το πακέτο των τσιγάρων ροζ και όμορφο, είναι σαν να λες τα κορίτσια είναι χαζά. Ε, εγώ ξεκίνησα να καπνίζω με κανονικά τσιγάρα και βλέποντας και τα πακέτα με τις προειδοποιήσεις που υπάρχουν. Γιατί ήδη απαγορεύεται τα, τα, τσιγάρα να κυκλοφορούν χωρίς τις προειδοποιήσεις εδώ και 18 χρόνια στη χώρα μου. Όποιο κατανοήσει ότι κάνει κακό στην υγεία, το τσιγάρο θα σταματήσει να καπνίζει. Έχω την εντύπωση ότι α, γυρνάμε γύρω από το θέμα χωρίς να μπαίνουμε στην ουσία. Δεν είναι το πακέτο ε, η ουσία του θέματος, είναι το περιεχόμενο. Έπειτα, σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα σε νοικοτήνη, είμαι και εγώ σε αυτήν την ακρόαση, αλλά πιστεύω ότι όταν διατίθεται στα φαρμακεία μπερδεύω τον καταναλωτή. Ουσιαστικά είναι σαν να παίρνουμε το εμπόριο από μια επιχείρηση και το δίνουμε σε μια άλλη. Πρέπει να είμαστε σοβαροί. Όταν ε, ο άνθρωπος αγοράζει κάτι από το φαρμακείο, το συνδέει με κάτι που είναι καλό για την υγεία. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ αυστηροί στην νομοθεσία και σε καμία περίπτωση να μην ε, διατίθεται στα φαρμακεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Χέπνερ, η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζουμε αυτό να είναι η βάση για την πρόταση της Κομισιόν. Συμφωνώ με τη Λίντα, πρέπει να έχουμε μια απαγόρευση διασυνοριακών πωλήσεων. Δεν θέλουμε δηλαδή να κάθεται οι άνθρωποι μπροστά στον υπολογιστή τους και να παραγγέλνουν τσιγάρα από το ίντερνετ. Τώρα, όσον αφορά αυτά που θα μπαίνουν πάνω στο πακέτο, ναι, χρειάζεται και εκείνα ρύθμιση. Δεν ε, πρέπει να υπάρχει καμία διακόσμηση για να τα κάνει πιο ελκυστικά αυτά τα πακέτα. Όπω είπε και η Λίντα, χρειάζεται μεν απαγόρευση. Πρέπει δεν να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούν να ε, δράσουν ω προ την ενημέρωση των ε, καταναλωτών και ενδεχομένως να, μπορούν, να πρέπει να υποχρεωθούν και οι εταιρείε να πληρώσουν για αυτή την ενημέρωση. Χρειαζόμαστε εκστρατείε ενημερωτικέ. Υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα καπνού για τα οποία πρέπει να ενημερωθούν οι καταναλωτέ, με τα οποία οι εταιρείε προσπαθούν να προσελκύσουν παιδιά στο κάπνισμα. Τώρα το προϊόν καθ' αυτό. Ναι, υπάρχουν όντω ορισμένα πρόσθετα τα οποία είναι σήματα, τα οποία χρησιμοποιούν μάλλον οι εταιρείε και τα πρόσθετα αυτά πολλές φορές είναι γεύσεις, γεύσεις που αλλοιώνουν την ε, πραγματική γεύση του καπνού και αυτές οι γεύσεις πολλές φορές είναι εθιστικές και εδώ πρέπει να επέμβουμε. Τώρα τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, αν μπορούσαμε καλό θα ήταν να ε, απαγορεύαμε να καπνίζει ο κόσμος ε, ηλεκτρονικά τσιγάρα σε δημόσιους χώρους διότι περιέχουν νοικοτήνη. Σε ορισμένε ε, χώρες μάλιστα έχει τεθεί ένα ελάχιστο όριο ηλικίας ε, που μπορεί κάποιο να καπνίσει τέτοιο τσιγάρο. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι κάτι που δεν είχα ακούσει μέχρι πριν από λίγου μήνε. και από τότε... Από τότε που άρχισα λοιπόν να ενημερώνομαι, είχα εκατοντάδες επιστολές από ανθρώπους που μίλησαν για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα υπερασπίστηκαν και μου είπαν δοκίμασα τα πάντα. Έχω δοκιμάσει τα νοικοτήνη, ετό, νατάλιο. Ξανά άρχισε το κάπνισμα. Όμω αυτά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα πραγματικά κάνουν δουλειά. Έχω σταματήσει να καπνίζω και είμαι απόλυτα πεπισμένο για την αξία του. Για την αξία του και ότι αυτά τα τσιγάρα αποτρέπουν τον κόσμο από το να πεθάνει από το τσιγάρο. Περιμένω ακόμα από την Κομισιόν να κάνει μια πρόταση ε, που θα περιορίζει την νοικοτήνη. Η πρόθεση της ε, Κομισιόν φυσικά δεν είναι να υποστηρίξει το ηλεκτρονικό τσιγάρο και να οδηγήσει με ε, περισσότερο κόσμο στην κατανάλωση νοικοτήνης. Έχω ένα, μια επιστολή από έναν καθηγητή ο οποίος λέει ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο για μένα είναι πραγματικά καταστροφικό κό καταστροφική εφεύρεση. Καταστροφική για ποιον όμως, για τις καπονοβιομηχανίες φυσικά, έτσι. Επίσης, μου γράφουν πολλοί ότι αν περάσεις κάποιο καιρό καπνίζοντας ηλεκτρονικό τσιγάρο, θα συνειδητοποιήσεις ότι το κανονικό τσιγάρο έχει αειδιαστική γεύση. Οι καπνιστέ λοιπόν, οι πρώην καπνιστέ, με το που αλλάζουν ε, προ το ηλεκτρονικό τσιγάρο, ανακαλύπτουν ότι ο καπνό όντω έχει απέσια γεύση. Και πιστεύω πραγματικά ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο μπορεί να σώσει ζωέ. Όλοι αυτό μου λένε. Και όσον αφορά τώρα του νέου και το πόσο ελκυστικό θα είναι, να σα πω ότι δεν νομίζω να φαίνεται κάποιο κουλ cool και ωραίο όταν καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο. Ένα έφηβο, ε, το αντίθετο μάλιστα. Φαίνεται γελίο αυτό το θέμα. Chris. Και μετά η κυρία Βέστελου. Eh, Μάλιστα, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Βρίσκω πολύ καλή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να, για να μειώσει το τσιγάρο. Η Λίντα έκανε μια πάρα πολύ καλή έκθεση και δεν περίμενα και τίποτα άλλο από εκείνη. Όμως πραγματικά να ε, μιλήσω και για το ζήτημα του σνούς. Θέλω να το θίξω πάλι. Κανεί φυσικά δεν υποστηρίζει ότι ο καπνό νου είναι κάτι ωφέλιμο, είναι κάτι χρήσιμο. Όμω η Σουηδία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτή την εξαίρεση, να μπορεί δηλαδή να συνεχίζει να πουλά αυτόν τον καπνό σνου. Και εάν δεν μπορεί πια να πουλήσει αυτόν τον καπνό, τότε η επιφύλαξη που είχε η Σουηδία, η εξαίρεση που έγινε σεβαστή όταν μπήκε η Σουηδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πλέον θα έχει καταστρατηγηθεί. Ο σνούς, καπνός είναι σνούς. Πρόσθετα ή όχι, είναι ένα σουηδικό προϊόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να μας πει εκείνη τι είναι, τι, τι μπαίνει, τι δεν μπαίνει. Σας παρακαλώ να εξαιρεθεί ο καπνός σνούς από αυτήν την οδηγία. Είναι ένα προϊόν το οποίο ρυθμίζεται με πάρα πολύ άσχημο τρόπο από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Σουηδία είναι η χώρα στην οποία κινείται αυτό το προϊόν και είναι η χώρα η οποία θα πρέπει να ρυθμίσει τις ε, διατάξεις με αυ... για αυτό το προϊόν. Και πραγματικά, εγώ προσωπικά θα προτιμούσα να μην αναφέρεται καθόλου αυτός ο καπνός στην οδηγία. Ε, Νομίζω ότι θα πρέπει να αποκλειστεί από το άρθρο 6 ο καπνός για τα οσνούς, για τα προσθετικά και τα, τις αρωματικές ουσίες γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί μόνο μερός η Ευρωπαϊκή Ένωση να ορίζει τι είναι αυτό ο καπνό νόσο και αν μπορούμε να τον χρησιμοποιούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Λύση είναι Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ τη Λίντα για την πρόταση εκθέσεω. Εγώ συμφωνώ με τη γραμμή την οποία εκπροσώπησε ο συγγητή τη Ομάδα μου, ο κύριο Καρλ Χάιντ Φλόρεντς. Την υποστηρίζω πλήρω. δεν θα τα επαναλάβω όλα. Δύο-τρία μόνο πράγματα για, τις, για τα πρόσθετα, για τις πρόσθετες ουσίες. Έγινε λόγος για, τον, για τη ζάχαρη, αναφέρθηκε και νωρίτερα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να ε, προσέξουμε το θέμα αυτό, διότι η επανεισαγωγή των ε, ειδικών επιδοτήσεων για τον καπνό ε, αποφασίστηκε από την Ολομέλεια, παρά τις αντιστάσεις κάποιων από εμά. Ελπίζω ότι δεν θα υποστηρίξει τίποτα σε αυτό το Συμβούλιο που ξέρουμε ότι δεν θέλει μέχρι στιγμή τουλάχιστον ειδικέ επιδοτήσει για τα προϊόντα καπνού. Ε, πιστεύω επίση ότι θα πρέπει ιδιαίτερα να, γίνει έμφαση, να δοθεί έμφαση στου κινδύνους του παθητικού καπνίσματο. Αναφορά λοιπόν προειδοποίησεως με εικόνα και με ε, γραπτή αναφορά για τους κινδύνους του παθητικού καπνίσματος πάνω στο η συσκευασία, θα ήταν κάτι πολύ σημαντικό, αλλά επίσης και το ξέρω αυτό από την καριέρα μου ως γιατρού, ότι μπορεί και πρέπει να το γράψουμε αυτό, να οδηγήσει και σε αποβολή το κάπνισμα και σε... και ε, σε άσθμα, παιδικό άσθμα. Αυτό ότι πρέπει να το λέμε γιατί χρειάζεται να υπάρχει αυτή η υπαγρύπνηση Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο ομιλητή, παρακαλώ. Ναι, θα είμαι σύντομο γιατί ήδη ακούστηκαν πολλά. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την τόσο ένθερμη, θέλετε και γλαφυρή παρουσία που μα έκανε. Αλλά θέλω να πω ότι η καταπολέμηση του καπνού και η ενημέρωση των νέων για να αποφύγουν να γίνουν καπνιστές Αυτό δεν γίνεται έτσι με τέτοιε απαγορεύσει και τέτοιου περιορισμού ώστε αναγκαστικά οι καταναλωτέ να μπουν σε μια συγκεκριμένη γραμμή. Αυτό αντίθετα μπορεί να γίνει καλύτερα με την μόρφωση και την κατάρτιση στα σχολεία και μέσω ειδικών ε, πρωτοβουλίων όπω έκαναν κάποιε χώρε, στη χώρα μου για παράδειγμα, απαγορεύεται η πώληση στους ανηλίκους ή απαγόρευση του καπνίσματος συγκεκριμένου χώρου. Το να μπαίνουμε τώρα σε τόσο σημαντικού τομεί. όπως η χρήση μιας απλής συσκευασία ε, χωρίς ε, μάρκα, χωρίς τίποτα. Ε, αυτό δεν και άλλα ζητήματα. Λειτουργία ιστορική αγορά, πνευματική ιδιοκτησία, ε, στρέβλωση του ανταγωνισμού. Επίσης, ε, ε, τα όρια σε κάποιες ουσίες χωρίς α, επιστημονικές αποδείξεις θέλω δεν έχει νόημα και πάλι αυτό μπορεί να ενισχύσει τον αθέμετο ανταγωνισμό. Αν εγκριθεί ε, η οδηγία α, έχει, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε αυτό το κακό αποτέλεσμα για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Συμφωνώ με την προηγούμενη παρέμβαση που είπε ο συνάδελφος ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο έχει σκοπό να μειώσει το κάπνισμα. Αν βάλουμε και άλλους περιορισμούς, αποθαρρύνουμε τον καπνιστή που προσπαθεί να μειώσει το τσιγάρο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σατατεβίλιο. Σας ευχαριστώ. Ακούσαμε πολλά διαφορετικά επιχειρήματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την συγγετρία και τους και που συνεργάστηκαν στην υπόθεση αυτή. Θα ήθελα να υπογραμμίσω μία πτυχή σχετική με το λαθρεμπόριο. Πολλοί μίλησαν ήδη για το λαθρεμπόριο τσιγάρων και θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς αξιολογεί ε, την κλίμακα στην οποία δεξάγεται το λαθρεμπόριο αυτό έχει προσμετρήσει το φαινόμενο αυτό. Λέγεται εν γέννη ότι 35% των προϊόντων καπνού στις αγορές μας είναι προϊόντα απομίμησης ή προέρχονται από πηγές ε, λαθρεμπορίου. Υπάρχουν ενδείξει ότι μπορεί να είναι και 50% ακόμη, να φτάσει στο 50% που στο το ποσοστό αυτό. Το θεωρεί ω ε, σημαντικό πρόβλημα αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάποιοι λένε ότι το ζήτημα είναι η φύλαξη των συνόρων. Εγώ που είμαι από τη Λιθουανία και έχουμε εξωτερικά σύνορα με, χώρες, με χώρα μη μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, θεωρούμε ότι χρειάζεται να εισαχθεί μια ειδική νομοθεσία. Δεν νομίζετε ότι πρέπει το επίπεδο του, το επίπεδο του να αυξηθεί αν δεν ενισχύσουμε τους ελέγχους. Μίλαν, να έχεις τον λόγο εσύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχάς να υπογραμμίσω ότι το κάπνισμα χωνεύει. Οδηγεί σε εθισμό, εξάρτηση και πρέπει να το βλέπουμε σε κάτι το κακό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είμαι πεπισμένο ότι κάποιο όμω θα αποφασίσει να σταματήσει το κάπνισμα μόνος του. Βεβαίω θα πρέπει να του δώσουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, τις σωστές και αληθεί πληροφορίες και να υποστηρίξουμε εκείνον ο οποίο θέλει να θεραπευθεί από αυτή την εξάρτηση. Ξέρουμε ότι πολύ συχνά αυτός που θέλει να σταματήσει το κάπνισμα χρειάζεται ε, βοήθεια από ειδικού για να βελτιώσει πιθανότητες του να καταφέρει να κόψει το κάπνισμα. Η εκπαίδευση επίση έχει, η παιδεία που δίνουμε στους νέους έχει επίδραση στο αν θα αρχίσει ένα νέο να καπνίσει. Τα δικά μου τα παιδιά παραδείγματα δεν καπνίσουν γιατί τα έχω έτσι αναθρέψει. Επίση, Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μπορούμε να αφήσουμε στην ε, καπνοβιομηχανία. Υπάρχουν πολλά άλλα θέματα τα οποία θα πρέπει να υπαρθούν στην ε, ε, αρχή της επικουρικότητας. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν μας από μια έκθεση να προτείνουμε κάθε δυνατό κανόνα ο οποίος θα ρυθμίζει τα πάντα. Ας ασχοληθούμε με τα ουσιώδη ζητήματα και ας αναλογιστούμε και τι σφάλματα έχουμε διαπράξει στο παρελθόν και τι είδους έθιμα, και τι είδους έθιμα έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο το κάτω. Ευχαριστώ κύριο Σχέρνερ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Το γεγονό ότι προσπαθούμε να αποτρέψουμε τους νέου να αρχίσουν το κάπνισμα είναι καλό, αλλά να δούμε γιατί τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς που ήδη καπνίζουν. Πιστεύω λοιπόν πως είναι μεγάλο λάθος να ρυθμίζουμε τα λιγότερο βλαβερά προϊόντα καπνού. Είναι μία λάθος, μία κακή ρυθμιστική πολιτική. Ο σνούς είναι ένας καπνός που δεν προκαλεί καπνό και να σας κάνω μια υποθετική ερώτηση. Τι θα, γίνει, εάν, τι θα γινόταν εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είχε απαγορεύσει το κρασί αλλά είχε επιτρέψει τη βότκα. Κάπως έτσι είναι αυτό τώρα με τον καπνό και το σνούς που λέτε. Δηλαδή απαγορεύοντας το κρασί στην Ευρώπη αλλά επιτρέποντας τη βότκα θα ήταν σαν ας πούμε να ρύθμιζε τα πάντα εκτός από το λευκό κρασί στη Γαλλία. Είναι ένα ε, προϊόν ο ΣΝΟΥΣ, που λέμε ότι δεν θέλουμε στην ε, εσωτερική αγορά. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Είτε θα τον δεχτούμε στην εσωτερική αγορά και θα τον ρυθμίσουμε καλά και αυστηρά, είτε θα πούμε όχι, δεν τον θέλουμε τον σνου στην εσωτερική αγορά και στην περίπτωση αυτή δεν τον ρυθμίσουμε καθόλου. Αλλά αυτή η παράνοια με τον σνου που λέμε ότι ναι, να τον απαγορεύσουμε στην Ευρώπη αλλά να τον ρυθμίζουμε στη Σουηδία είναι περίεργη, είναι αδιανόητα, τα κατανόητα και πραγματικά συμφωνώ με την προσέγγιση του Chris Davidson, δηλαδή πια που είπε ότι να κάνουμε ότι ό,τι αποτρέπει τους ανθρώπους να καπνίσουν καλό και να συμφωνήσουμε τουλάχιστον στο ε, αν το θέλουμε ή δεν το θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όχι να πούμε ότι ναι, δεν τον θέλουμε μεν στην ενιαία αγορά, αλλά να τον ρυθμίσουμε στη Σουηδία. Όχι. Επόμενο ε, ομιλητή, ο κύριος Κουμουτσάκος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, καλωσορίζω την ε, πρόταση οδηγίας ε, και την δουλειά που έχει κάνει η συνάδελφος για τα προϊόντα καπνού. Βεβαίως στόχος είναι η προστασία των νέων μας από την εθιστική συνήθεια του καπνίσματος. Και πιστεύω ότι η πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί από την εισηγήτρια της Επιτροπής μας έχουν αυτό στόχο και ορθώς κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα όμως να εκφράσω έντονο προβληματισμό μου ως προς ειδικά ένα σημείο και λόγω του περιορισμένου χρόνου. Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν και θα, αν υπάρχουν θα ήθελα να τα γνωρίζω. Επαρκή ερευνητικά δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι τα τσιγάρα τύπου slim είναι περισσότερο ελκυστικά για τους νέους πριν αρχίσουν το κάπνισμα ενώ όλοι ξέρουμε ότι καταναλώνται από μεγαλύτερη ηλικία χρήστε. ήδη χρήστε. Ας μην ξεχνάμε ε, άλλωστε ότι το μέτρο της κατάργησης των SLIM δεν είχε περιληφθεί στο προσχέδιο του κειμένου τη Επιτροπή. Δεν είχε περιληφθεί. Και δεν έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Επομένως θεωρώ ότι η συγκεκριμένη κάθετη και χωρίς καμία εξαίρεση ή ευελιξία απαγόρευση που προτείνεται στις τροπολογίες ε, της ε, συναδέλφου έχει ένα υψηλό ποσοστό αυθαιρεσίας. Κατά τα λοιπά υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία θα μπορούσε κανείς να συζητήσει. Γενικά η κατεύθυνση είναι σωστή, αλλά ειδικά αυτό το θέμα νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ε, πολύ. Επόμενος ομιλητή, ο κύριο Κυλακάκης. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον, την εισηγήτρια. Προσωπικά δεν έχω κάνει ούτε ένα τσιγάρο στη ζωή μου. Ούτε μία φορά. Δεν ξέρω λοιπόν τι χάνω. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι στις αρχές της δεκαετίας του 70 μου είπαν πολλά και είχα πάρα πολύ καλές πληροφορίες έτσι ώστε να μην αρχίσω το κάπνισμα. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω στην αξία της πληροφόρηση. Έχει να κάνει με τη στάση μας, με τον πολιτισμό μας και με το πόσο φτηνό ή ακριβό είναι το προϊόν του καπνού και πώς επιτρέπεται και πόσο μάλλον επιτρέπεται να το καπνίσεις μέσα στο σπίτι ή έξω από αυτό. Τώρα όταν προσπαθούμε να κάνουμε το κάπνισμα αγαθό. Δεν είμαι σίγουρος εάν είναι η σωστή προσέγγιση, διότι χαμηλώνοντας την τιμή θα δώσουμε ένα πλεονέκτημα στα λαθρέα τσιγάρα και αυτό θα κάνει πιο εύκολο το να αρχίσουν οι νέοι το κάπνισμα ε, και ιδιαίτερα στο νότο της Ευρώπης το πόσα χρήματα έχεις είναι καθοριστικό για το αν θα αγοράσει ή όχι τσιγάρα. Αν δεν έχεις δεν παίρνεις. Άκουσα ότι είπατε για τις προσπάθειες να σταματήσουμε τους νέους να αρχίσουν το κάπνισμα και εγώ πιστεύω όμως αντίθετα ότι προσπαθούμε να μειώσουμε το ποσοστό των νέων που θα αρχίσει. Υπάρχουν πολλοί νέοι που καπνίζουν και που δεν πρόκειται να το κόψουν. Συμφωνώ με τον Κρίς και με οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια έχει αναφερθεί για να βοηθήσει τους καπνιστές. Μιλάμε για μια μεγάλη πλειοψηφία ανθρώπων που θα επηρεαστούν. Αυτοί οι ίδιοι οι καπνιστές. Θα ήθελα λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να δούμε τα πράγματα λαμβάνοντας υπόψη και τους καπνιστές. Ο Μάριο Πρίλιον, ο επόμενος ομιλητής. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το κάπνισμα κάνει κακό. Είμαι πρώην καπνιστής για 25 περίπου χρόνια. Και για αυτό το λόγο ακριβώς κάνω ό,τι μπορώ για να μειωθεί η βλάβη στην υγεία από το καπνό. Η εισηγήτρια μας έδωσε μια σειρά από στοιχεία που είναι ανησυχητικά πρέπει λοιπόν να υπάρχει καλύτερη πρόληψη για την υγεία, για να μειωθεί το κοινωνικό κόστος, την ιατρική περίθαλψη και τα, άρα και το οικονομικό κόστος που συνεπάγεται το κάπνισμα. Βλέπουμε τώρα μια σειρά προτάσεων που αφορούν κυρίως η συσκευασία. Κυρίως για να, να πιστούν οι νέοι και οι γυναίκες. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τεχνάσματα για να πείσουμε τους νέους. Ο βασικός στόχος είναι η προστασία της υγείας του πολίτη. Μια ναι, υγεία πραγματικά α, τίθεται σημαντικό κίνδυνο από α, τους ανενδύαστους πολιτές και κατασκευαστές. Αν δεν είναι το κόστος των σιγάρων, αν δεν είναι το προβλήματα στην υγεία που δημιουργεί το κάπνισμα. Τι άλλο μπορείς να κάνεις, τι άλλο μπορείς να πεις για να μειώσεις ε, τη βλάβη που προκαλεί το κάπνισμα. Εγώ εστιάζω πιο πολύ στην πρόληψη. Με στοχευμένες πρωτοβουλίες που να φοβίζουν τους ανθρώπους α, για τις συνέπειες του καπνίσματος μόνιμες ασθένειες που απαιτούν πολύ δαπανηρές και επώδυνες θεραπείες. Αν καταφέρουμε να πείσουμε τους ανθρώπους ότι πρέπει να μειωθεί σημαντικά το κάπνισμα και να δημιουργήσουμε νέες γενιές που δεν καπνίζουν, τότε θα έχουμε κάνει πολύ σημαντική δουλειά και θα έχουμε προστατεύσει και την οικονομία μας ταυτόχρονα. Θα εξετάσω τις τροπολογίες και πιστεύω ότι θα υποβάλω και εγώ κάποιες δικές μου. Ο πρόεδρος ε, διέκοψε τον ομιλητή, λέει ότι δεν έχουμε ακόμη χρόνο, έχουμε πολλούς ομιλητές στον κατάλογο. Μπορείτε να παραλάβετε, λέει ο ομιλητής. Ε, πρέπει να περάσω στον επόμενο ομιλητή, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ. Λοιπόν, στον κατάλογό μου, ε, στρέκεται μαζί. Ε, ο and next speaker is please. Uh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στην έκθεση αυτή η Λίντα. Συμφωνώ στα όσα λέει για τις ε, τυποποιημένες συσκευασίες είχαμε ακούσει διάφορα παράδοξα ότι η τυποποιημένη διαδικασία θα προσελκύει ακόμη περισσότερο στο κάπνισμα του νέου, γιατί θα μετατρέψει τη συσκευασία σε απαγορευμένο καπνό και δεν ξέρω τι. Δεν καταλαβαίνω αυτά τα επιχειρήματα, ούτε καταλαβαίνω γιατί μπορεί κανείς να καταλήξει τι συμπεράσματα. Για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι δύσκολο το θέμα, πολύ λόμπινγκ έχουμε υποστεί και καταλαβαίνω ότι βοηθάει κάποιου ενδεχομένω ή νομίζουν ότι του βοηθάει για να σταματήσουν, αν βοηθάει έστω, αλλά χρειάζεται να ρυθμιστούν τα ηλεκτρονικά αυτά τσιγάρα. Και αν είναι ε, ε, ε, φαρμακευτικού τύπου το, το προϊόν αυτό, έτσι θα πρέπει να ρυθμιστεί. Και πάντως δεν θέλουμε να απαγορευτούν, γιατί αν βοηθάνε κάποιον να κόψει το τσιγάρο είναι πάρα πολύ καλό. Πρέπει όμως να εξασφαλιστεί μια μακρύτερη περίοδος ε, προσαρμογής έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ε, απρόσκοπτη ολοκλήρωση προς διαδικασίες της αδειοδότησης. Εγώ θα ήθελα να ακούσω τα επιχειρήματα όλων των πλευρών πριν καταλήξουμε στο αν θα, αλλά πάντως δεν νομίζω ότι θα πρέπει να απαγορευτούν. Ε, πάντως Νομίζω ότι κάποιες συνελφοί μερικές φορές παρασύρονται όταν μιλάνε για τα ηλεκτρονικά σιγαρέτα. Για τον Αργιλέ νομίζω ότι δεν αληθεύει ότι τον χρησιμοποιούν μόνο πιο ηλικιωμένοι. Εγώ έχω ακούσει, πίσω, κάνω λάθος, ότι φαίνεται πολύ μοντέρνος και cool κάποιος νέος που καπνίζει την αργυλέ ε, την σημερινή ημέρα. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που λένε ότι πρέπει να προσέξουμε την επιπλέον προσθήκη ζάχαρης αλλά και την αμμονία που καθιστά πάρα πολύ εθιστικά τα σιγαρέτα. Ευχαριστώ πολύ, Εστέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κι εγώ έχω υπάρξει καπνίστρια, ευτυχώς. Δυστυχώς, α, αναγκάστηκα να γίνω και μάρτυρας του θανάτου φίλων μου που πέθαναν από καρκίνο που συνδέεται με το κάπνισμα. Είναι γνωστό ότι το κάπνισμα σκοτώνει, κάνει κακό στην υγεία και υποστηρίζω την της προτάσει, αλλά θέλω πιο πολύ να επισημάνω το εξή μια εξαιρετική περίπτωση, μια ιδιαιτερότητα που δεν έχει να κάνει ούτε με ελκυστικό περιτύλιγμα, ούτε με την γκλάμορ εμφάνιση, ούτε την προστασία της υγείας του πολίτη, που είναι και τα πρωτεύοντα. Αναφέρω κάτι άλλο, κάτι που αφορά το εξή. Ίσως λόγω άγνοιας δεν έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι τεχνικές πτυχές της συσκευασίας που ισχύουν σε κάποιες χώρες. Πιο συγκεκριμένα μιλώ για τις διαστάσεις της συσκευασία που χρησιμοποιείται ε, σε μια περιοχή της Πορτογαλίας ε, στις Αζόρες που είναι πιο μικρά ε, πακέτα. Δεν έχω σκοπό να προσεγγίσω κανένα. Απλά είναι πιο μικρά τα τσιγάρα, πιο μικρή συσκευασία. Αυτό λοιπόν που λέει το 13. Ότι είναι δυνατόν τα, τα πακέτα να είναι από χαρτί ή από άλλο σκληρό υλικό και μετά στο άρθρο 9, στο G, λέει το κείμενο ότι το ύψος δεν μπορεί να πάνω από 64 χιλιοστά και το εύρος όχι πάνω από 95 χιλιοστά. Αυτές οι συσκευασίε που σας δείχνω δεν εμπίπτουν σε αυτές τις διαστάσεις. Αυτά τα εργοστάσια που κατασκευάζουν τα τσιγάρα και που έχουν μια ζωή πάνω από 100 ε, χρόνια, που κάνουν αυτή την υπηρεσία, καταλαβαίνετε τι σημαίνει για θέσει εργασία κτλ. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, πρέπει να μου δώσετε τρία λεπτά. Περιμένω τόσο ώρα να μιλήσω και θα μου δώσω τον χρόνο να εκφράσω την άποψή μου. Ιδίω μιλώ για μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση. Πρόεδρος, ναι, οι άλλοι όμως ήταν σκιώδεις ηγητές και γι' αυτό είχαν προσθέτω χρόνο ως σκιώδεις ηγητές. Όταν ξεπερνάει κανείς τα 2,5 λεπτά, ανακαστικά τους δεκόπτω, σας καταλάβαμε για το μέγεθος της συσκευασίας. Όχι, όχι, μα δεν είναι αλήθεια. Λοιπόν, θεωρώ ότι και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Γιατί το να βάλουν λουκέτο αυτά τα εργοστάσια σημαίνει ανεργία που ήδη είναι πολύ ψηλή στη χώρα μου και οικονομικές συνέπειες πολύ οδυνηρές. Τώρα δεν μιλάμε μόνο για προστασία υγεία, αλλά μιλάμε για σεβασμό μιας ιδιαιτερότητας ε, σε μια χώρα όπως η Πορτογαλία. Ε, η κυρία Ριβαζή, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Λίντα για την έκθεση αυτή προσφέρει πολλές λύσεις. Εγώ νομίζω ότι πρέπει πάρα πολύ να ξέρουμε τι θέλουμε. Στόχος μας είναι να μειώσουμε τον αριθμό των καπνιστών. Δύο είναι οι κύριες πτυχές αν προκειμένου. Η ελκυστικότητα αφενός ή εξάρτηση αφετέρου. Ελκυστικότητα. Εδώ βεβαίως έχει σημασία η συσκευασία. Εγώ σας έφερα φωτογραφίες όπου ακριβώς ε, επιλέγεται μια συσκευασία για γυναίκες και θυμίζει είτε ένα κραγιόν είτε μια συσκευασία ε, make-up λοιπά. Είναι αυτό που ονομάζεται sexy, δηλαδή θεωρεί μια γυναίκα ότι εντάξει καλό είναι αυτό να το έχω στο τσαντάκι μου, δεν μπορεί να βλάπτει. Ε, εδώ λοιπόν είναι το ζήτημα της ε, συσκευασίας πολύ σημαντικό, γιατί αν βάλουμε μια φωτογραφία καρκίνου των πνευμόνων ή καρκίνου του λάριγκα, αν και δεν θέλω να φτάσω μέχρι εκεί, νομίζω ότι κόβουμε την, την όρεξη. Επιπλέον, ε, γιατί όλα αυτά τα αρωματικά, βανίλια, σοκολάτα και φρούτα, γιατί να κόψουμε αυτή την πικρή ταγκιά γεύση του καπνού. Ε, εμείς ακριβώς αυτό λέμε, ότι πρέπει να περιορίσουμε στο μέγιστο δυνατό την ελκυστικότητα του καπνού για τον νέο. Και επίσης, αυτό το οποίο δεν συστήκα αρκετά, είναι η εξάρτηση. Η νοικοτήνη μεν προξενεί από μόνη της εξάρτηση. Αλλά είναι όλα αυτά τα πρόσθετα και εγώ θα ήθελα να έχουμε έναν θετικό κατάλογο που να πούμε τι επιτρέπεται να έχει μέσα αποκλειστικά το τσιγάρο. Ξέρω πολύ καλά ότι με τους αρνητικούς καταλόγους ε, η καπνοβιομηχανία, όπως άλλωστε και η φάρμακοβιομηχανία, θα, κάνει, θα, θα βρει τον πλάγιο δρόμο και θα, θα βγάλει λίγο από μια ουσία, θα προσθέσει λίγο από μια άλλη και θα πει, κοιτάξτε, είναι νέα ουσία, δεν προβλέπεται στο αρνητικό κατάλογο. Ε, η αμμονία, η αμμονία διευκολύνει την μετά μετάβαση της νοικοτήνης στον εγκέφαλο. Γι' αυτό ενισχύει την εξάρτηση. Εάν λοιπόν τα απαγορεύσουμε αυτά θα μειωθεί η εξάρτηση και για το ηλεκτρονικό τσιγάρο το τελευταίο. Εγώ συμφωνώ έστω Εάν υπάρχουν αυτά τα τσιγάρα θα πρέπει να είναι φαρμακευτικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα από αυτό που σημαίνει. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρία Σχάλντομούζα. Θα είμαι σύντομη. Υποστηρίζω την πολύ ε, κομψή και καλή προσέγγιση της Λίντα. Νομίζω ότι και η ε, εικόνα και η ε, διαστάσεις μία της συσκευασία έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Εγώ, ε, χωρίς να είμαι καπνίστρια, όταν είδα τέτοιου είδους συσκευασίε για γυναίκες, όπως λέμε, girly, πρέπει να ομολογήσω ότι είχα όρεξη να τις φέρω στο χέρι μου, να τις δω, να τις γυρίσω προς πίσω, να τις κοιτάξω. Ε, αυτό λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ομοθεσία μας. Χαίρομαι που έχουμε την ε, ακρόαση για το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Έχω ακούσει και εγώ πολλά πράγματα γι' αυτό. Καλό είναι να ανταλλάξουμε πληροφορίες, να συλλέξουμε υλικό, να δούμε τι είναι καλό σε αυτήν την υπόθεση, τι δεν είναι. Πρέπει να ρυθμιστούν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα με μια νομοθεσία που δεν θα είναι απαγορευτική, αλλά που θα ρυθμίζει και θα ε, δίνει την έμφαση στην απαλλαγή από την εξάρτηση στον καπνό. Εν τέλει δε, η οδηγία για το καπνό και τα προϊόντα του στόχο έχει να μειώσει την εξάρτηση από τα προϊόντα καπνού των νέων, αλλά πρέπει να καλύπτει και αυτούς που ήδη έχουν αρχίσει να καπνίζουν και είναι εξαρτημένοι. Άρα πρέπει να δούμε και τα θέματα του κινδύνου στα ε, λεγόμενα συνήθη κοινά προϊόντα καπνού, δηλαδή τα ποστά της πίσας, ε, εκεί που δεν υπάρχουν πρόσθετες ουσίες. Ε, αυτά όμως που αποτελούν κίνδυνο για την υγεία του καπνιστή. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Οκονή. Ευχαριστώ πολύ Λίντα και συγχαρητήρια για την έκθεση, αλλά πρέπει να πω ότι μένω άναυδιος προς ένα-δύο πράγματα. Ο Κάλς Φρόνς έχει φύγει μένα, αλλά συχνά λέει ότι είναι πρόβλημα δημόσιας υγείας το κάπνισμα και βεβαίως με 300 νεκρούς το χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα την ημέρα προφανώς εννοεί η ομιλήτρια, είναι σαν να πέφτει κάθε μέρα ένα αεροπλάνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα αν έπεφτε ένα αεροπλάνο κάθε μέρα στου ευρωπαϊκού ουρανού, θα απογορεύαμε την κυκλοφορία, την ενέργεια κυκλοφορία. Άρα πρέπει να πάψουμε πια να υποκύπτουμε σε αυτή την ε, πίεση που ασκεί με όλη τη δύναμη η καπνοβιομηχανία. Για τι φωτογραφίε και τι εικόνε πάνω στα ε, πακέτα των τσιγάρων. Και αυτά γκέρλι και γυναικεία πακέτα συμφωνώ απολύτω πρέπει να απογραφθούν. Για τι φωτογραφίε, εγώ δεν βλέπω κανένα πρόβλημα. Γιατί δεν είναι η λύση το 65, το 75% κτλ. Υπάρχουν επιχειρήσεις, μάρκε μάρκες ρούχων για νέους, ε, για ε, αξεσουάρ γυναικεία κτλ. Οι οποίες φτιάχνουν ε, ε, πακέτα τσιγάρων μοδάτα με πολύ ωραία διακόσμηση μέχρι και με νεκροκεφαλές στολισμένες με διαμαντάκια τα οποία προβλέπονται για να μπει μέσα το κανονικό πακέτο τσιγάρων που είχε αγοράσει κανείς στο περίπτερο. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια διαφορετική λύση και πάνω απ' όλα η ε, παιδαγωγική λύση πρέπει να λειτουργήσει. Η ανατροφή, η ε, παιδεία στα σχολεία, από το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, αλλά και, και διαφημιστικά σποτ, την ώρα που κάθεται κανείς να φάει διαφημίσεις από τις δημόσιες υπηρεσίες, από τα Υπουργεία Υγείας ή οτιδήποτε άλλο, διαφημιστική ή εκστρατεία που θα δείχνει την ώρα που κάθεται η οικογένεια για φαγητό μαζί, τι είδους συνέπειες μπορεί να έχει ο καπνός. Και επίσης το κόστος, το κόστος έχει πολύ μεγάλη σημασία για το αν θα έχει πρόσβαση ο νέος στο τσιγάρο ή όχι. Πρέπει να είναι όλες οι χώρες στην, ε, στην ίδια τιμή και να είναι πολύ ψηλή αυτή η τιμή και πρέπει να σας πω ότι είμαι πρώην καπνίστρια. Ο πρόεδρος, ε, συγχαίρω όλους αυτούς που ήταν πρώην καπνιστές, βλέπω ότι είστε πολλοί εδώ οι παρόντες και συγχαρητήρια που καταφέρατε να το κόψετε. Και τελευταίος ο μηνυτής, ο κύριος Μιλοσάτσης. Ευχαριστώ πολύ Κάιλ. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να κλείσω με μια διαφορετική νότα αυτή τη συζήτηση. Βλέπουμε τα πράγματα από οικονομική σκοπιά. Και πραγματικά αυτές τις μέρες το μόνο που καταλαβαίνουμε είναι το χρήμα. Όμως είναι καθήκον μας να δείξουμε στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς, πόσο κοστίζει, αφού λοιπόν όλοι σκεφτόμαστε με βάση το χρήμα, πόσο κοστίζει ένας ασθενής που πάσχει από χρόνιο άσθημα, ο οποίος χρειάζεται ιατρική φροντίδα χρόνια. Πόσα λεφτά κοστίζει λοιπόν αυτό ο ασθετής από το, στο κράτος. Πόσα λεφτά κοστίζει ένας ασθενής με καρκίνο του πνεύμονα, με, όλου, με όλες τις ασθένειες που προκαλεί το κάπνισμα. Αυτό πρέπει να τους δείξουμε, διότι κοστίζουν τόσα χρήματα λοιπόν στο κράτος και στο τέλος πεθαίνουν κιόλας. Αυτοί οι ασθενείς δεν πηγαίνουν στη δουλειά και αντί να πάνε στη δουλειά πρέπει λοιπόν να πάνε στο νοσοκομείο, να υποστούν ε, την ε, περίθαλψη, την αγωγή και το κράτος χάνει χρήμα. Αυτές τις, ε, μου φαίνεται πως αυτές τις μέρες δεν, κανέναν δεν αγγίζει ο, αν, ο άνθρωπος, το ανθρώπινο στοιχείο. Όλοι ενδιαφέρονται για το χρήμα. Το χρήμα κινεί τα πάντα αν κάνουμε αυτό θα εξοικονομήσουμε τόσα χρήματα στο σύστημα υγείας και από την άλλη θα εξοικονομήσουμε... θα γλιτώσουμε και πολλού πολίτε μα. Ε, πραγματικά με σοκάρει το γεγονό ότι συναδέλφοι από άλλε επιτροπέ έρχονται σε αυτήν εδώ την επιτροπή ε, ω εμπειρογνώμονε και πιστεύουν ορισμένοι από την άλλη ότι αυτό το πρόβλημα δεν είναι τόσο σοβαρό. με την ψήφο σας θα παραλύσετε τις προσπάθειες που κάνουμε προς τους πολίτες και αυτό με λυπεί. Δεν είμαι αδιάφορος γι' αυτό. Ξέρετε ότι όλο ένα και περισσότεροι νέοι άνθρωποι, 14, 15 χρονών, αρχίζουν το κάπνισμα, νέα κορίτσια. Είναι επιδημία. Ως άνθρωπος και ως γιατρός πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πάρα, πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και θα επιδεινωθεί διότι αυτές οι γυναίκες αργότερα θα γίνουν μητέρες και όταν θα μείνουν έγκυες Ευχαριστώ πολύ, διέκοψε ο Πρόεδρος, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρω ότι είστε τρεις. Θα μοιράσετε λοιπόν μεταξύ σας το χρόνο. Και μετά θα ολοκληρώσουμε. Πέντε λεπτά λοιπόν στο τέλος χρόνο για τη Λίντα και αρχίζετε. Ευχαριστώ για το λόγο. Θα μιλήσω εξ ονόματο και των συναδέλφων. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε την εισηγήτρια για την εξαιρετική έκθεση, όπω και όλου του κοιόδη και του άλλου αξιότιμου ευρωβουλευτέ για τα σχόλια και τι ερωτήσει. Φυσικά με χαρά σημειώνουμε το γεγονό ότι η εισηγήτρια υποστηρίζει πολλά από τα μέτρα που προτείναμε κι εμεί, οπότε θα εστιάσω την παρέμβασή μου εκεί όπου βλέπουμε μία απόσταση στι απόψει μα. Πρώτα απ' όλα, η απλή συσκευασία. Και εμεί το εξετάσαμε το ενδεχόμενο αντί για πλήρω τυποποιημένη συσκευασία. Το μελετήσαμε στην πληκτική όμω καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι σε αυτή τη φάση μια τέτοια μερική προσέγγιση θα ήταν ε, καλύτερη. Γιατί? Για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα, κείμενη οδηγία δεν απαιτεί προειδοποιήσεις με εικονογραφήματα. Μόνο 10 κρατημέλη το κάνουν αυτό. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι μεγαλύτερε υποχρεωτικέ εικονογραφήσει ω προειδοποιήσει είναι το επόμενο σημαντικό βήμα. Δεύτερον, είναι πολύ μικρή η εμπειρία ε, που έχουμε από την τυπομημένη συσκευασία. Μόλις στην Αυστραλία γίνεται αυτό ακόμη. Οπότε πρέπει να δούμε πόσο αποτελεσματική είναι αυτή η τακτική αυτή η προσέγγιση σε σχέση με την δική μας πρόταση βεβαίως ε, σημειώνουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση κέρδισε μία δίκη στο Νότο Αυστραλινό Δικαστήριο αλλά επειδή ακόμα δεν έχετε δικήσει, περιμένουμε να δούμε το τελικό νομικό καθώς κατά πόσον μπορεί να περάσει σε... και πρέπει να το δούμε σε λίγα χρόνια. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη από εκεί και πέρα να ε, θεσπίσουν πιο αυστηρά μέτρα των κρίνων αναγκαίων σύμφωνα με τη συνθήκη και επίση και εμείς δεσμόμαστε σε πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία ενσωμάτωσης ώστε να δώσω μια εικόνα για την εμπειρία που έχουμε κερδίσει ε, σε σχέση με αυτή την ε, ε, νέα συσκευασία σε ό,τι αφορά το δυσυνοριακό εμπόριο εξετάσαμε διάφορε εναλλακτικέ στη μελέτη και θεωρούμε ότι αυτό προτείνουμε υποχρεωτική κοινοποίηση για του λιανοπολιτέ που κάνουν ε, τηλεπολίσει συνειδητικά ώστε να έχουν έναν μηχανισμό ε, έγκριση ε, επαλήθευση είναι κάτι σημαντικό. Όμω καταγράφουμε και τα επιχειρήματα από το Κοινοβούλιο και από άλλου που λένε ότι αυτή δεν είναι κατάλληλη λύση. Σε ό,τι αφορά τα τσιγάρα σλιμ ε, ε, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτά τα προϊόντα είναι πιο ελκυστικά και στοχεύουν ιδίω στις γυναίκε και κυρίω στις κοπέλε. Αυτό το λένε και τα ίδια τα ιστορικά έγγραφα τη βιομηχανία. Θέλετε μια απόδειξη? Να βλέπετε ότι μπορείτε να πάρετε και δωρεάν δείγματα τέτοιων ζυγάρων από ένα website από τι μεγαλύτερε εταιρείε που παράγουν τα τσιγάρα. Αρκεί να δηλώσετε σε γυναίκα. Να λοιπόν, μια ξεκάθαρη απόδειξη ότι μιλάμε για marketing καθαρά Εντάξει, σε πιστεύουν. Λες σε άνθρωπο 18, το λες, σε πιστεύουν. Έτσι και σου τα δίνουν δωρεάν. Σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, πολλοί αναφέρθηκαν σε αυτό. Θέλω πρώτα απ' όλα να επισημάνω ότι η πρόθεσή μα δεν είναι να απαγορεύσουμε τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Γιατί κάποιοι αυτό είπαν. Αυτό που θέλουμε πρώτα απ' όλα, να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα α, δίνουν πλήρη δυναμικό ε, ε, ε, σε επίπεδο αισθήσεων και να μην χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση ως μία πύλη εισόδου των νέων στη χρήση της νοικοτήνης που είναι θεστική. Πολλά από αυτά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που χρησιμοποιούνται σήμερα δεν έχουν περάσει ούτε από έκρηση ούτε από αξιολόγηση και κάποιοι παρασκευαστέ ομολογούν ότι δεν μπορούν καν να εγγυηθούν το επίπεδο περιεκτικότητα σε νοικοτήνη. Αυτό είναι πολύ συγκεκριτικό. Δεν υπάρχει λοιπόν ίσω ανταγωνισμό ανάμεσα σε ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν νοικοτήνη και άλλε εναλλακτικέ ε, παραγωγέ που αντικαθιστούν την νοικοτήνη και έχουν εγκριθεί σε διάφορα κρατημέλη. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα επίση συχνά χρησιμοποιούνται ακριβώ για να δώσουν, ε, για να οδηγήσουν στην σταδιακή πάυση του καπνίσματο. Αλλά τελικά θα μπορούσε να πει κανεί ότι αν τελικά λειτουργούν τόσο καλά δεν θα υπάρχει πρόβλημα με την αδειοδότησή του. Κάποιο άλλο ζήτημα που ακούστηκε. Χαρακτηρισμό των συστατικών. Εμείς κυρίως εστιάζουμε στην ελκυστικότητα του προϊόντος. Θέλουμε να αποφύγουμε οι νέοι να ακολουθήσουν αυτή τη συνήθεια και νέοι σε πολύ νεαρή ηλικία να ξεκινούν να καπνίζουν. Και αυτά τα συστατικά είναι πολύ εύκολο να το πείσουμε, γιατί έχουν ένα και μόνο σκοπό που χρησιμοποιούνται. Μπορεί κανείς να παρασκευάσει τσιγάρα χωρίς τέτοιες αρωματικές ύλες και όταν χρησιμοποιούνται, χρησιμοποιούνται σε μεγάλες ποσότητες. Εμείς θέλουμε να δημιουργηθούν ε, πάνελ δοκιμών που να χρησιμοποιούν την οσμή και τη γεύση για να ε, αταξιολογούν. Από εκεί πέρα το λαθρεμπόριο των τσιγαρών ήδη υπάρχει και σε μεγάλο ποσοστό ε, και άρα ε, το να αναφέρεται η μάρκα του, του, τσιγάρου δεν ήταν πρόβλημα και όσο πιο ελκυστική και γνωστή είναι μια μάρκα τόσο πιο πολύ προσελκύει ε, τους απομιμητές. Άρα λοιπόν αυτή είναι η απάντησή μα. Θέλουμε να εστιάσουμε στο να κάνουμε ένα λιγότερο ελκυστικό προϊόν και να δώσουμε πιο πολλά μέσα στα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν το εθρεμπόριο. Επίσης, μια άλλη διάταξη τη πρότασή μα, και δεν να την επισημάνω, λέει ότι οι ουσίε που είναι γνωστές αποδεδειγμένα ότι ε, αυξάνουν τοξικότητα και τον εθισμό, θα απαγορευτούν. Α, ήδη κάποια κράτη-μέλη έχουν προχωρήσει και όσοι έχουν αποδεικνά στοιχεία είναι πολύ χρήσιμα για να μπορούμε να εμπνεύσουμε καλύτερα αυτή τη διάταξη. Τέλος, λίγα λόγια για του νους. Η κείμενη νομοθεσία ήδη ρυθμίσει για το σνούς. Απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση το σνούς. Η Σουηδία έχει μια παρέκκληση για μια πτυχή που είναι απαγόρευση ε, στη θέση στην εμπορία. Όλες οι υπόλοιπε πτυχέ ήδη ρυθμίζονται. Όλα λοιπόν για την να κτλ. Ε, ισχύουν για το σνούς. Αυτό είναι το status quo και δεν καταλαβαίνουμε εμεί στην Κομισιόν για ποιο λόγο να αλλάξει το status quo διότι δεν προτείνουμε καμία αλλαγή ουσιαστικά. Απλά θέλω να το εξηγήσω. Και τέλος, το τελευταίο σχόλιο. Πολλοί μίλησαν για σύγκρουση με τη θρονομαδασία, ιδίω με τα παιδί του ΠΟΕ. Είμαστε πεπισμένοι ότι η πρότασή μα είναι άδεια απόλυτα με του κανόνε του ΠΟΕ. Δεν δημιουργεί διακρίση η πρόταση αυτή. Σε καμία περίπτωση δεν δίνουμε πρόκλημα στου εγχώριου ε, ε παρασκευαστέ και αυτή η πρόταση έχει περάσει και το τεστ Σε Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ Λίντα. Θέλεις εσύ να ολοκληρώσει σύντομα, Πρόεδρε. Δεν θα απαντήσω σε όλες τις παρατηρήσεις. Γιατί θα μα φάει πολλή ώρα και έχουν οι διερμηνείς περάσει από τις 3 το απόγευμα και όλες τις ψηφοφορίες και όλα αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ του συναδέλφους για τη συμβολή τους. Από τα όσα λέτε, αντιλαμβάνομαι ότι θα εξασφαλίσουμε καλή νομοθεσία για τον καπνό, με κάποιες διαφορές βεβαίως που πάντα υπάρχουν. Για το ηλεκτρονικό σιγαρέτο θα κάνουμε το εργαστηριό μας. Κάποιοι βέβαια είπαν ότι είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις που το παράγουν. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι προς τώρα ηλεκτρονικά τσιγάρα προέρχονται από την Κίνα. Δεν προέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να είναι σαφές, γιατί είναι και ζήτημα Πρέπει να έχει κανείς ύψης της ποιότητας προϊόντα για να παραγάγει τέτοιου είδους σιγαρέτα. Δεν είναι λοιπόν μικρομεσαίες οι επιχειρήσεις, είναι εταιρείε ε, μεγάλου κυβισμού, πολλών εκατομμυρίων λιρών ε, στο, σε κεφάλαιο. Γι' αυτό δεν θέλω να έρχονται οι διάφοροι ε, καουμπόιδες και να εισάγουν στην αγορά σιγάρετα ηλεκτρονικά χωρίς ε, τεχνικές προδιαγραφές. Αυτό είναι κάτι λοιπόν το οποίο παρακολουθούμε. Ξέρουμε ότι και οι Ηνωμένε Πολιτείε παρακολουθούν το ίδιο θέμα. Η κυρία Κορνή έφυγε, αλλά ε, έχω στοιχεία να τη δώσω για το τι είδου ε, επίδραση μπορεί να έχει, ιδιαίτερα στον νέο καπνιστή, υποψήφιο καπνιστή, μια φωτογραφία που δείχνει αυτές τις ε, εικόνας. Βεβαίως αυτό δεν μπορεί να γίνει πάνω σε ένα μικρό πακετάκι το οποίο μοιάζει με πακέτο ε, αρώματος γιατί δεν έχει και το χώρο να μπει σχετική φωτογραφία. Για τα όσα είπε η κυρία τα τεχνικά, μικρά ζητήματα, μπορεί να καταθέσει τροπολογίες. Αλλά θα ήθελα να πω ότι το σημαντικό είναι ότι πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον το 5% επί της συσκευασία προειδοποίηση για να είναι ορατή στον ε, πολίτη. Όταν κάποιοι λένε ναι, χρειάζεται ενημέρωση του κοινού, συμφωνώ, ενημέρωση του κοινού για τα σιγαρέτα, αλλά δεν είναι δουλειά της, ε, των δημοσίων αρχών να το πράξουν αυτό. Είναι υποχρέωση της ε, ε Δεν μπορεί να πληρώνει το κράτος για αυτά, όπως υπόθηκε πολύ σωστά. Κάποιοι άλλοι είπαν ότι μπορούμε να βοηθήσουμε να πληρώνουμε δηλαδή ε, να προβλέψουμε τέτοιου είδους διεθνιστικέ ε, εκστρατείες. Μα κοιτάξτε όμως η όταν κάνει, όταν κάνει ε, διαφήμιση περνάει μοντέλα και ιδέες. είδα σε μια σκηνή στο Στρασβούργο την, μια γυναίκα μπροστά μου που περίμενε για να αγοράσει ένα πακέτο slim. Ήρθε η σειρά της λοιπόν, ζήτησε τα slim, η περιπτερούχο τη είπε: Α, δεν έχουμε αυτά τα τσιγάρα, αλλά πάρτε τα άλλα. Και αυτή επέμεινε λέγοντα: Όχι, όχι, αυτά είναι τα light. Εγώ αυτά θέλω. Επειδή ήταν slim, θεωρούσα ότι είναι light. Εδώ λοιπόν βρίσκεται όλη η παρεξήγηση, εδώ βρίσκεται όλη η, ε, ε η εσφαλμένη παρουσίαση της ε, αλήθειας με τα εκατομμύρια που ρίχνουν ε, οι εταιρείε καπνού. Ελπίζω λοιπόν με τη συνεργασία σας να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια καλή ε, νομοθεσία για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την ε, συμμετοχή και τη συνεργασία. 8 Μαΐου προθεσμία για την κατάσταση των τροπολογίων, 12 το μεσημέρι. Παρακαλώ μην καταθέτετε όμως όλη τελευταία στιγμή της ε, τροπολογία σας, γιατί αλλιώ τις άλλες ε, ημερομηνίες 29-30 για την ανταλλαγή ε, απόψεων για τις τροπολογίες και 11-12 12 Ιουλίου για την Επιτροπή για να δούμε πότε θα γίνει η ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Αύριο το πρωί 9 με συντονιστές. Χαίρετε.